πρέπει να παραστεί σε μια κηδεία στο Βερολίνο. Ελπίζουμε να μπορέσει να έρθει. Στη συνέχεια. Θα αλλάξουμε λοιπόν λίγο την μέτρια διάταξη. Στο Στρασβούργο συνεδρίσαν οι πολιτικές ομάδες. και πρότειναν σε ό,τι αφορά το σημείο 9 να διαγραφεί από την ημέρησια διάταξη για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Αυτό το θέμα λοιπόν αναβάλλεται για μια προσεχή συνεδρίαση. Άρα η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα γίνει το Μάρτιο δεν μας δημιουργεί εμάς πρόβλημα η αναβολή της έκθεσης αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν. Θα αναβάλουμε την ψηφοφορία για τον Οκτώβριο, 26-27 Οκτωβρίου. Συμφωνεί η συγγετρία βλέπω. Άρα δεν υπάρχει αντίρρηση, θα το αναβάλουμε. Εγκρίνεται λοιπόν η μερική διάταξη με τις τροποποίησεις αυτές. Τώρα, έχετε στο φακελό σας τα πρακτικά για τις 13-14 Ιουλίου και για τις, ε, για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για σχέδιο των πρακτικών μέχρι στιγμής ω ήθιστε. Αν δηλαδή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης τη Επιτροπής μας δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σημείο 3 ανακοινώσει του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα μεταδίδεται στο διαδίκτυο με έχω και εικόνα η σημερινή μας συνεδρίαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, είναι γνωστά. Δηλαδή, δεν υπάρχει διερμηνία για βουλγαρικά, τσέχικα, πορτογαλικά, σουηδικά, εσθονικά, λιθουανικά, λετονικά, σλοβενικά και μαλτέζικα. Σε όλες τις άλλες γλώσσες υπάρχει δηλαδή. Στα δανέζικα επίσης μπορείτε με να μιλήσετε αλλά όχι να ακούσετε διερμηνία από τα δανέζικα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διερμηνία. Όλα καλά, ωραία. Περάμε λοιπόν στο σημείο 4. Πρωτοβουλία πολιτών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο προκαλεί και μεγάλες συζητήσεις. Η κυρία Φοντούν η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα μας παρουσιάσει την πρότασή τη μετά την πρόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εν λόγω πρωτοβουλία. Γνωρίζετε ότι με βάση τη Λισαβόνα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ε, την ε, νομοθεσία, τη σύνταξη νομοθετημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ε, μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένε πρωτοβουλίε ο πολίτη και να δώσει συνέχεια σε αυτέ τι αιτήσει του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζονται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες από διάφορα κράτη-μέλη, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεούται να αναλάβει δράση, βέβαια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τις εκχωρούνται από τη συνθήκη. Και φυσικά σε σχέση με ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πολίτες. Και το οποίο φυσικά και έχει να κάνει με τις κοινοτικές αρμοδιότητες. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την πρωτοβουλία των πολιτών. για να ληφθεί δράση πρέπει να υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και ουσιαστικά να υπάρχει ένας κανονισμός και περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς αυτό συζητάμε. Έχουμε λοιπόν την απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο της ΑΦΚΟ, της Επιτροπής ΑΦΚΟ, αλλά γνωρίζετε ότι πρέπει επίσης και εμείς από δική μας πλευρά να προβούμε στις δέουσες ενέργειες. Ο Αλέν Λαμασούρ ορίστηκε ως εισηγητής με την Ζήτα έχουν ε, καταθέσει κοινό κείμενο οι δύο εισηγητές. Στις 8 Νοεμβρίου θα υποβληθεί στην Επιτροπή το κείμενο αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, προθεσμίες για την κατάσταση των τροπολογιών, Οκτωβρίου, άρα ψηφοφορία 27 Οκτωβρίου. 1 Οκτωβρίου λοιπόν για τις τροπολογίες σας και 27 για την ψηφοφορία. Στρέφομαι στην κυρία Φαντούν τώρα και μετά θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδεχομένως να έχει κάτι να μας πει. Κυρία Φαντούν, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, για την εισαγωγή που κάνατε. Μετά την ανάγνωση και την συζήτηση με εσά με τους την ανάγνωση του σχεδίου κανονισμού που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσα μια γνωμοδότηση για το νομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτών την οποία έχετε λάβει. Θα ήθελα λίγο σύντομα να μιλήσω για τα κύρια σημεία και για το πνεύμα της ε, γνωμοδότησής μου. Για να καταλήξουμε ελπίζω σε ένα θετικό συμπέρασμα έτσι ώστε η Επιτροπή μας να έχει θετική επιρροή στο τελικό έγγραφο και να το καταστήσουμε χρήσιμο και εύχριστο για τους ε, πολίτες. Ένα έγγραφο το οποίο θα βελτιώσει ίσως την ευρωπαϊκή νομοθεσία και οπωσδήποτε θα αναζωογονήσει τη συζήτηση για την Ευρώπη και θα φέρει την, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες και ταυτόχρονα ένα έγγραφο το οποίο θα είναι λογικό και δεν θα προκαλέσει πλημμυρίδα πρωτοβουλειών ε, οι οποίες θα προκαλέσουν ε, πρόβλημα στην Κομισιόν. Οπότε χρειαζόμαστε ένα απλό, λογικό έγγραφο, φιλικό όπως σας είπα προς το χρήστη και ταυτόχρονα ένα έγγραφο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα είναι η αρμόδια, θα μπορεί να λειτουργήσει κιόλας. Για μένα λοιπόν το βασικό θέμα όσον αφορά το έγγραφο αυτό και ε, τα όσα αναφέρω στην γνωμοδότησή μου ήταν το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για μια οργανωτική επιτροπή. Ένα φορέα ο οποίο θα συγκεντρώνει τι υπογραφέ. Μιλάει επίση, μιλάει λοιπόν η Κομισιόν για μια οργανωτική επιτροπή εγώ κάνω λόγο, μιλάνε για τους οργανωτές. Εγώ μιλάω για την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από φυσικά πρόσωπα. Είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Οπότε, όπως το βλέπω εγώ και ελπίζω να συμφωνείτε, η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τα φυσικά αυτά πρόσωπα. Ε, συζητήθηκε το από πόσε χώρες πρέπει να προέρχονται. Εγώ προτείνω 9 χώρες, το 1 τρίτο των κρατών μελών φυσικά πρόσωπα από το 1 τρίτο των κρατών μελών. Και προτείνω να είναι πολίτες που δεν έχουν άλλο τρόπο να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα ερετή πολιτική. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εγγραφή και το αποδεκτόν του πράγματος. Εδώ πέρα διαφέρω από την Κομισιόν. Η Κομισιόν πρότεινε κάποια πράγματα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους κοιόδης οι οποίοι ήταν θετικοί και έχω την εντύπωση πως όλοι συμφωνούμε στην πρόταση πως ε, τα άτομα που θα αποτελούν την Οργανωτική Επιτροπή δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγράψουν αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά να μαζέψουν υπογραφές και μετά να τους απαντήσει η Κομισιόν ε, για το παραδεκτό ή όχι. Η εγγραφή και το παραδεκτό του αντικειμένου πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι ένας ενίος έλεγχος, μία πράξη για αυτούς που κάνουν την έτσι. Ταυτόχρονα η Κομισιόν πριν την ε, τελική απόφαση για το παραδεκτό πρέπει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για το ποιο νομικό μέσο θα είναι το καταλληλότερο για την εκάστοτε πρωτοβουλία. Μπορεί να είναι οδηγία, κανονισμός, σύσταση. People who will gather later the million, one million of signatures should know what they aim at. Um,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 Πάω λίγο πίσω, λέει ο μιλητή. Εάν κάνετε ένα λεπτάκι προς τα πίσω, κύριε του. Συνεχίστε, παρακαλώ. Πού είχαμε μείνει, ναι, η Οργανωτική Επιτροπή την οποία προτείνω αποτελείται από φυσικά πρόσωπα από εννέα χώρες, οπότε θα συγκεντρώσει το 1 εκατομμύριο αυτό υπογραφών και την ε, δήλωση στήριξη. Θα υπάρχει λοιπόν ένα έντυπο με τα δεδομένα των ανθρώπων που έχουν υπογράψει. Προτείνω έναν ελάχιστο αριθμό δεδομένων. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία και χρόνος γέννησης και υπογραφή για μένα αυτά αρκούν. Με τους σκιώδεις ε, συζητήσαμε το εάν είναι απαραίτητος ο αριθμός ταυτότητας ή άλλων γράφων. Νομίζω πως δεν είναι απαραίτητος. Και επίσης το έγγραφο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ε, μικρότερο, για λόγους που ξέρετε. Αν κατάλαβα καλά δηλαδή, το έγγραφο το οποίο προτείνει η Κομισιόν αποτελείται από 6 σελίδες. Εάν δηλαδή έχουμε 6 εκατομμύρια σελίδες για να τι φέρει κάποιο στην Κομισιόν, ε, δεν είναι και τόσο καλό και για τα δάση. Προτείνω λοιπόν ένα μικρό έντυπο, μικρή προώθηση μέσω του διαδικτύου και ελάχιστα δεδομένα. Όνομα, τόπος και χρόνος γέννησης, ε, διεύθυνση, υπογραφή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στο έντυπο αυτό είναι πληροφορίες για την οικονομική στήριξη. Χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια για τις πηγές χρηματοδότησης αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Και εδώ πέρα συμφωνήσαμε πλήρως με τους κοιοδησίγητες. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και εγώ στην στην τροπολογία το έχω θέσει ξεκάθαρα, πως θα πρέπει να υπάρχει μια εκστρατεία πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και θα πρέπει να ενημερωθούν ε, οι πολίτες για το πώς μπορούν να οργανώσουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα που μπορούν να ενημερώσουν τους πολίτες, όπως το Νεολαία σε δράση, το Europe Direct, όλα αυτά τα γραφεία πληροφόρησης που υπάρχουν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσωπείες της Κομισιόν οι πολίτες ε, πρέπει να έχουν ε, σωστές πληροφορίες για το ποια θέματα είναι παραδεκτά για να οργανωθούν, για να μην κάνουν ε, πάρα πολλά λάθη, για να μην απορρίψει τις προτάσεις η Κομισιόν και μετά να αποθαρρύνονται και να ασκούν κριτική στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ποιοι λοιπόν θα οργανώνουν και ποιοι θα υπογράφουν. Η πρότασή μου είναι πως η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε ηλικία η οποία τους επιτρέπει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Αλλά το, οι άνθρωποι οι οποίοι υπογράφουν το ένα αυτό εκατομμύριο, όπως ξέρετε, στις ε, εκλογές περισσότερες χώρες ε, είναι και στην οποία μπορεί να ψηφίσει κανείς 18, αλλά στην Αυστρία είναι 16 παραδείγματο χάρη. Οπότε προτείνω να είναι εκεί και το κατόφλι, να επιτρέψουμε στους 16χρονους να υπογράφουν και εάν η παρενέργεια, αν θέλετε, αυτού είναι να έχουμε και μια δυναμική ευρωπαϊκή συζήτηση, θα είναι κάτι το θετικό αυτό, το να συμπεριλάβουμε δηλαδή τους νέους. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της ε, γνωμοδότησής μου και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας και αναμένω την ε, επικοδομητική συνεργασία μαζί σας για να έχουν οι πολίτες ε, ένα μέσο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ σαφή αυτή παρουσίαση. Παρουσίαση που μας δίνει και μια πολύ καλή βάση συζήτησης. Πριν όμως περάσουμε στη συζήτηση. Ναι, παρακαλώ. Να το ξαναπώ. Όχι, ας ακούσουμε πρώτα τους βουλευτές και μετά να ακούσουμε την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ ξεκάθαρη έκθεσή τη. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την έκθεση και καμιά δυο ερωτήσει επί τη ουσία. Δεν ξέρω βέβαια αν ε, μπορούμε να τι θέσουμε αυτέ σήμερα τι ερωτήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενημερωτική εκστρατεία προ όλου του Ευρωπαίου πολίτε, θέλω να ρωτήσω το εξή. Ποιο θα χρηματοδοτεί στην ενημερωτική αυτή εκστρατεία, Ένα άλλο πράγμα περιορισμός στον αριθμό των ερωτήσεων σε αυτή την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Και επίσης ε, η τελική ψηφοφορία έχει κάποια νομική ε, αξία, δηλαδή αν ψηφιστεί και δεν γίνει αποδεκτή μια πρωτοβουλία, έχει κάποια νομική αξία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απλά πρόκειται για μια σύσταση. Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Kiitoksia sitten Rova Saahe ja sen... Ευχαριστώ πολύ. Sorry, my name sounds different in Finnish. I couldn't recognize... Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα ότι είπατε το όνομά μου στα φιλανδικά, κύριε Πρόεδρε. Δεν το αναγνώρισα όπω το προφέρατε, αλλά δεν πειράζει. <laughs> Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια. Ε, την εισηγήτρια είναι πολύ ε, καλή η έκθεση και είναι και πολύ σημαντικό και εμείς να συνεργαστούμε σοβαρά για αυτό το θέμα. Είναι καλό για του πολίτε. Έχω μια ερώτηση για το διαδίκτυο την πτυχή αυτή της πρωτοβουλίας των πολιτών, διότι όπως αναγνωρίσατε και εσείς, η όλη διαδικασία της υποβολής μιας πρωτοβουλίας πολιτών θα οδηγεί σε ενδεχόμενα ή θα ενισχύσει, θα προωθήσει τις συζητήσεις. Παρότι ε, μπορεί κάποιες φορές να μην φτάνει το εκατομμύριο ο αριθμός των υπογραφών. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας χώρος στο διαδίκτυο, ένα είδος φόρουμ, όπου θα μπορούσαν οι πολίτες να συζητούν τα διάφορα ζητήματα. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο των νέων μέσων ενημέρωση, είπατε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ασφαλέ περιβάλλον για τη συλλογή υπογραφών και στήριξης, υποστήριξης. Ίσως θα ήταν δύσκολο για τα μεμονωμένα άτομα να διασφαλίσουν ότι η συλλογή των υπογραφών γίνεται με ασφαλή τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν μήπως υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματο χάρη, να έχουμε κάποιο λογισμικό ανοιχτή πηγής, open source, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι πολίτε αν θέλουν να, να δρομολογήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών. Και επίσης το θέμα της πρόσβασης στις πληροφορίες σε σχέση με τις ε, ενδεχόμενες πρωτοβουλίε πολιτών, αν θα μπορούσε ε, να υπάρχει, αν θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση δηλαδή των πληροφοριών και αν αυτό θα μπορούσε να γίνει εύκολα, αν η αναζήτηση δηλαδή θα μπορούσε να είναι εύκολη. Και αν αυτή η πτυχή της ενημέρωσης θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα ε, στην οποία γίνεται και η κατάθεση των πρωτοβουλειών ε, πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σκαβαντάχη τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι οι δύο συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα έκαναν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία υπογραμμίσατε. Ε, Καταρχάς, εννέα χώρες μου φαίνεται μία διάσταση πάρα πολύ λογική για να ε, πετύχουμε το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Συμφωνώ μαζί σας ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή οργανωτική, γιατί θα πρέπει να δώσουμε μία κάποια μορφή στο όλο θέμα. Τώρα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ενδεχόμενα από πού ε, και πώς θα δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή και το κοινοβούλιο είναι μια καλή είναι ένας ε, μπορεί, πρέπει να έχει έναν ρόλο καθοδηγητικό και δεν θα είναι η εκτελεστική επιτροπή που θα πρέπει ε, να συμμετέχει ε, γιατί αυτοί θα πρέπει να δράσουν αφού συγκεντρώσουν τον αριθμό των υπογραφών. Απ' την άλλη πλευρά θεωρώ ότι είσαστε πάρα πολύ σωστή όταν ε, λέτε ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε και όσον αφορά τον αριθμό των πληροφοριών που θα δίνουν ε, οι πολίτες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Επίσης ε, για, την, τα, για, την, για τον εντοπισμό των χρηματοδοτήσεων δεν θα μου έκανε εντύπωση οι, τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη, να, να, να αναλάβουν συγγνώμη, ε, την χρηματοδότηση. Στο, μιλάμε ε, για μια πρωτοβουλία η οποία δεν θα πρέπει να καθοδικηθεί από τα διάφορα λόμπι, θα πρέπει να είναι κάπως ε, ανεξάρτητη οικονομικά. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη να αναλάβουν τα απαραίτητα ε, οικονομικά μέσα ε, για να χρηματοδοτηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η πρωτοβουλία των πολιτών, γιατί στο κατω ε, γιατί δεν μιλάμε για πολλά χρήματα. Τώρα όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία, σαν βουλευτής δεν ξέρω δεν μπορώ να παρέμβω στην, ε, στην νομοθεσία των κρατών μελών. Άλλα κράτη θεωρούν ε, ότι η ενηλικίωση γίνεται στα 16 χρόνια, άλλα στα 18. Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια παράλληλη ε, νομοθεσία. Μπορούμε απλούστατα να πούμε ότι για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα δημοψήφισμα η νόμιμη ηλικία είναι η ηλικία η οποία προβλέπεται από την νομοθεσία κάθε κράτου μέλους. Επίσης ε, ε, υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουμε 6 εκατομμύρια σελίδες, διότι μία... Ε, ένα κείμενο τέτοιο, τέτοιας μορφής θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα ή δύο σελίδες το πολύ και όχι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κουτσουρέψουμε τα κοινοτικά τα, τα δάση γενικότερα για να κάνουμε τέτοιου είδους ψηφίσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καβαντά. Θα απαντήσει η συγγήτρια και μετά θα περάσουμε στις επόμενες τρι, τρεις ερωτήσεις. Ε, είναι δύσκολο να διαβάσω, είναι πολύ δύσκολο να διαβάσω τα ονόματά σας από εδώ, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη εκ των, προτέρων για, την, ε, για το πώς προφέρω τα ονόματά σας. Κυρία Τούνου. Ε, input. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα, θα χρηματοδοτήσει την εκστρατεία δεν διευκρινίζεται στο κείμενο και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες, διότι καταρχάς ε, δεν έχουμε εμπειρία για το πόσο θα οργανωθεί το θέμα. Επίσης υπάρχει και, το, και η αναθεώρηση, το ενδεχόμενο αναθεώρησης ε, μετά από εμπειρία τριών ετών. Και μετά θα πρέπει να, να δούμε αν θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο ή όχι. Εάν το όργανο αυτό χρησιμοποιείται συχνά, θα πρέπει να το δούμε αυτό πρώτα. Τώρα ποιος θα χρηματοδοτήσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η διαφάνεια. Κάποιες όμως εκστρατείες μπορεί να είναι ακριβές, κάποιες όλες όμως όχι με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Χρειαζόμαστε τόσο πολλά χρήματα, δηλαδή μπορεί οι οργανωτές να χρησιμοποιήσουν και χορηγούς και ποιο θα είναι το ποσό δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει, ότι θα πρέπει να νομοθετήσουμε εξαρτάται από τα θέματα. Άλλα θέματα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, για άλλα θέματα οι οργανωτές θα, θα οργανώνουν πιο μεγάλη εκστρατεία. Το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η απόλυτη διαφάνεια. Αυτό ενδιαφέρει πιστεύω. Κατά τα λοιπά, δεν πρέπει να ρυθμίσουμε νομοθετικά το θέμα της χρηματοδότησης και δεν το ρυθμίσουμε στο κείμενο. Τώρα όσον αφορά το ίντερνετ, πιστεύω ότι είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα ε, να ε, προωθήσουμε την ε, συλλογή υπογραφών, συγκέντρωση υπογραφών μέσα από το ίντερνετ. Ούτως ή άλλως θέλουμε να έχουμε μια απλή και ασφαλή χρήση του ίντερνετ και για τα θέματα αυτά. Και αυτό θα μπορούσε να ε, αποτελέσει και μια παρενέργεια ε, τη πρωτοβουλία των πολιτών στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή ότι το ίντερνετ τελικά θα παίξει έναν πιο αποτελεσματικό ρόλο. Εξού και υπέβαλα αυτή την τροπολογία ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συγκέντρωση υπογραφών μέσω του ίντερνετ. Διότι αυτό δεν πατάγει σε όλες τις γλώσσες, συγγνώμη, σε όλε τι χώρε, όπω ξέρετε. Ε, δεν θέλουμε να συνεχίζουμε να κόβουμε δέντρα και να καταστρέφουμε δάση, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τι υπογραφέ μέσω του ίντερνετ. Και συμφωνώ απόλυτα. Δεν δίνω μια συνταγή, δεν ξέρω κάποια συνταγή για να προωθήσουμε τη συγκέντρωση υπογραφών μέσω του ίντερνετ. Εγώ λέω ότι απλώς πρέπει να το κάνουμε. Το ίδιο και για τις πηγές χρηματοδότησης που θα πρέπει να εμφανίζονται στο ίντερνετ. Τώρα, έτσι όπως περιγράφεται το όλο θέμα στο κείμενο, η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει μια πλατφόρμα πληροφοριών. Πρόκειται για ε, πρωτοβουλία πολιτών. Επομένως, οι πολιτές θα ενημερώσουν, οι πολίτες θα βρουν πηγές πληροφοριών και οι πολίτες ε, που συγκεντρώνουν τις υπογραφές θα οργανώσουν και αυτή την πλατφόρμα ε, ενημέρωσης και, για την, ε, και θα πρέπει τα κράτη απλώς να επιτρέπουν να υπάρχει ε, δυνατότητα υπογραφής ενός τέτοιου κειμένου στο ίντερνετ. Με, ασφαλές, με ασφαλή τρόπο. Ναι, ναι, λέει η κυρία Φοντούνα. Αυτό εξαρτάται όμως από το πώς λειτουργεί το ίντερνετ και διαφέρει από κράτος σε κράτος. Τώρα, για το κράτος ε, που θα πρέπει να αναλάβει τις, ε, ε, τα την χρηματοδότηση. Νομίζω ότι απάντησα. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολιτών, άρα δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε στο κράτος. Τα, οι πολίτες θα πρέπει να οργανώνουν τη χρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν, σας, δεν σας κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά για να είναι τα πάντα διάφανα θα πρέπει τα κράτη να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση. Ας πούμε, όταν ψηφίζετε στη χώρα σας, ε, δεν πληρώνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, το κράτος πληρώνει τις εκλογές. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με αυτό το δημοψήφισμα. Πρόκειται για ένα δημόσιο, δημόσια διαβούλευση και θα πρέπει το κράτος να πληρώνει, για να μην έχουμε τα λόμπι. Δεν το συμπεριέλαβα αυτό στην τροπολογία μου, λέει η κυρία Φοντούν, γιατί δεν πρόκειται για πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Είναι μια πρόταση για την υιοθέτηση ε, κάποιου ομοθετικού κειμένου. Λοιπόν, είναι ε, μια πρόταση για την... Ούτως ή άλλως μιλάμε για, ε, για την ηλικία, μιλάμε για πάνω από 18 ετών. Λοιπόν, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από χορηγούς, από διάφορες δραστηριότητες ε, πολιτών κτλ. Επομένως, δεν πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ότι εμείς που ενημερώνουμε τους ψηφοφόρους μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή ότι σε, αυτή την, σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να διευκολύνουμε τη συγκέντρωση των υπογραφών. Δεν είναι εκλογές, δεν μιλάμε για ένα, για ένα κείμενο μυθιστικού περιεχομένου. Είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν το συμπεριέλαβα. Και για μένα πρόκειται για μια ξεχωριστή δράση από τις εκλογές. Γι' αυτό και ο ρόλος του κράτους είναι διαφορετικός στην περίπτωση αυτή. Έτσι πως το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Αλλά είμαι ανοιχτή και σε περαιτέρω συζητήσεις. Επίσης συζητήσαμε για την ελάχιστη ηλικία, την ομιλικία. Τι άλλο, υπήρχε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι απήντησα. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση υπόσχεται πολλά εάν συνεχίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε, ίσως αυτό οφείλεται και στην ποιότητα της εισηγήτριάς μας και την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ε, συναντήσεις ε, που οργάνωσε και για το τι μας άκουγε. εξ ονόματος της ομάδας μου θα πρέπει να εκφράσω την συμφωνία μας με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προτάσεών της για τη διαφάνεια, κυρίως για αυτό το άνοιγμα όσον αφορά τον, τα διάφορα sites ε, των πολιτών, για την απλούστευση αλλά και την ε, ανάγκη να προστατεύσουμε και τους πολίτες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν όμως και κάποιες απορίες ακόμα, κάποια ερωτηματικά. Κυρίως όσον αφορά την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από φυσικά πρόσωπα μόνο. Κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες ε, ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουμε την Επιτροπή αυτή στους πάντες και να δώσουμε την δυνατότητα να γίνει ένα όργανο των λόμπι αλλά πιστεύω ότι οι μη κερδοσκοπικές ε, οργανώσεις, που είναι οργανώσεις πολιτών, θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο εδώ. Είχαμε μία συζήτηση με την εισηγήτρια σε αυτό το θέμα. Ε, δεν ικανοποιήθηκα πλήρως, οφείλω να ομολογήσω και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ζητήσουμε περαιτέρω, γιατί δεν πιστεύω ότι τα φυσικά πρόσωπα από μόνα τους έχουν την ικανότητα να α, υλοποιήσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τώρα, όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Καβαντά, με το κάνουμε και συνήθεια βέβαια, ε, αυτό το θέμα της δημόσιας χρηματοδότησης είναι κάτι το οποίο και εμείς το συζητήσαμε δεν είναι απλά τα θέματα, γιατί όλοι θέλουμε να αποφύγουμε τα λόμπι παντός είδους. Οι πολίτες από μόνοι τους διερωτώμεθα πού θα βρουν τα χρήματα. Εμείς στην συνεδρίαση ε, των σκιώδων εισηγητών είχαμε μιλήσει για κοινοτική χρηματοδότηση. Αλλά είχαμε πει ότι ε, εάν ε, ζητήσουμε την κοινοτική χρηματοδότηση, η Κομισιόν θα είναι και διάδικος και κατηγορούμενος, ε, και δικαστής και διάδικος. Ε, επομένως, ε, θα πρέπει στα θέματα του αποδεκτού να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κομισιό έχει μία τάση να περιορίζει τις πρωτοβουλίες, διότι ακριβώς πρόκειται για την Κομισιό που θα παίξει το ρόλο και δικαστή και διάδικου. Επίσης, Εκτιμώ ιδιαίτερα το ανοιχτό μυαλό της εισηγήτριας να συμπεριλάβουμε και τους νέους. Δεν θα πρέπει να το μπερδέψουμε αυτό με το δικαίωμα ε, συμμετοχής στις εκλογές, ε, διότι εδώ είναι άλλο θέμα. Μιλάμε για την ε, διευκόλυνση πρόσβασης στα θέματα της ηθαγένειας και του πολίτη. Ούτως ή άλλως μιλάμε για άτομα τα οποία θέλουμε να εντάξουμε στην κοινωνία μας, για άτομα τα οποία ζουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα με ένα νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης θεωρώ πως ε, συμφωνούμε ή μπορούμε να συμφωνήσουμε πως η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία των πολιτών ε, θα είναι επιτυχημένη μόνο εάν τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Και από την άλλη βεβαίως ε, αν διασφαλίσουμε πως δεν θα γίνει και τίποτα το περίεργο με την συλλογή των υπογραφών. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια λογική ισορροπία μεταξύ της λιγότερης γραφειοκρατίας, αλλά για να μην υπάρχει και απογοήτευση, αλλά να διασφαλίσουμε βεβαίως πως οι κατάλογοι των υπογραφών που θα κατατίθενται πράγματι θα είναι πραγματικές υπογραφές. Αλλά συμφωνώ με την άποψή σας πως αυτό το οποίο χρειαζόμαστε ως δεδομένα για την υπογραφή πρέπει να είναι ως το δυνατόν λιγότερα. Νομίζω και εγώ πως επαρκούν αυτά τα οποία είπατε. Όνομα, επώνυμο, τόπος κατοικίας γέννησης και ημερομηνία γέννησης και υπογραφή. Νομίζω πως αυτά επαρκούν για να ταυτοποιηθεί ένα άτομο. Οτιδήποτε άλλο νομίζω παρά είναι. Και... Είναι πράγματα τα οποία βέβαια γίνονται όχι μόνο και στο ίντερνετ, αλλά και από τη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, ε, από όπου κατάγουμε υπάρχουν ε, τέτοιες ε, πρωτοβουλίες που μαζεύουν υπογραφές στους ε, δρόμους και άμα τους δάνε υπογραφές τα παρατάνε και λένε πού να ψάχνουν τώρα τον αριθμό ταυτότητας και πρέπει πράγματι λοιπόν να αρκούν αυτά τα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά το διαδίκτυο θεωρώ πως πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις δυνατότητες αλλά όπως σας είπα να υπάρχει κάποια μορφή ηλεκτρονικής υπογραφής για να διασφαλίσουμε πως όντως το άτομο το οποίο υπέγραψε ταυτοποιείται για να μην υπάρχει καμία κατάχρηση για να διασφαλίσουμε πως πράγματι και εδώ πέρα έχουν κατατεθεί πραγματικές υπογραφές όσον αφορά τη χρηματοδότηση θεωρώ πως είναι κάπως δύσκολο το πρόβλημα, γιατί εάν είναι να είναι επιτυχής αυτή η πρωτοβουλία, τότε βεβαίως δεν είναι δυνατόν μόνο οι οργανώσεις εκείνες μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν να καταθέτουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος τότε που περιγράψει η κυρία Βερζιά, ότι μόνο λόμπι θα έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία και να μαζέψουν ένα εκατομμύριο υπογραφές στην Ευρώπη. Γιατί βεβαίως αυτό προϋποθέτει πως θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαφήμιση με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα είναι μόνο λόμπι που θα μπορούν να ξεκινήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά και απλοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν μεγάλα μέσα στη διάθεσή τους. Ξέρω πως αυτό ισχύει και για τις πρωτοβουλίε που έχουμε στην ε, πατρίδα μου, οπότε υπάρχει η δυνατότητα δωρεών για να χρηματοδοτηθεί η διαφημιστική καμπάνια. Θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε για τα νομικά πρόσωπα ε, να γίνει μια διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων αφενός ε, και κοινοφελών ενώσεων από την άλλη, αλλά αυτό θα είναι δύσκολο. Γιατί πού βρίσκεται το όριο. Και αυτό δεν είναι σωστό λοιπόν. Οπότε νομίζω πως ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις για το πώς θα διασφαλίσουμε πως δεν θα εκμεταλλεύονται αυτό το μέσο μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εάν θέλουμε πραγματικά να είναι ένα μέσο το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες της Ευρώπης και θα δημιουργήσουμε άλλη μία απογοήτευση ε, στους πολίτες και θα λένε «Ε, αυτά είναι για όσους έχουν λεφτά. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή και ο λόγος ε, των πολιτών και η συζήτηση στο τι κάνει η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Αν συμφωνείτε, Καλά θα να μιλήσει και ο αντιπρόεδρος μας, ε, γιατί μετά θα φύγει και στη συνέχεια θα δώσω στους υπόλοιπους συναδέλφους ε, που έχουν ζητήσει το λόγο. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι θα λάβετε το λόγο. Αν συμφωνείτε να προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούσαμε να μιλήσω στα δανέζικα, είπατε κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Άρα θα συνεχίσω στα δανέζικα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Φοντών για την έκθεση αυτή. Την έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω πως έχει ενσωματώσει αρκετά από τα στοιχεία που αναφέραμε ήδη. Και ε, δεν μπορεί... Πράγματι, σωστό είναι αυτό το οποίο είπατε να περιορίζονται τα στοιχεία σε μια σελίδα και όχι σε 6-7 και όχι μόνο για τα δέντρα όπως είπατε. Όπως ξέρετε άμα βλέπει κανένα πάκο ο πολίτης αρχίσει να λακίζει. Οπότε, όπως ε, και κάποιοι άλλοι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία μου έκαναν ε, εντύπωση αρνητική δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορούμε να λέμε πως κάποια κράτη-μέλη έχουν το όριο ηλικία στα 18, οπότε θα πρέπει να το κατεβάσουν ε, στα 16. Εντάξει, να το συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε μετά πώς θα, ε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω, εκτός αν σας παρεξήγησα, εγώ Προσωπικώς ε, ανησυχώ λίγο για αυτά τα 16 έτη τα οποία είπατε. Μετά το ερώτημα για το τι θα γίνει εάν κατέβει η ηλικία στα 16. Θα έχει όντως αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο είπατε. Ευχαριστώ τον λόγο. Τώρα έχει η κυρία Ζεράλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν τσέχικα σήμερα, θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω κυρία Τούν για το έργο της ε, και για την συζήτηση με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Άγγιξε νομίζω όλα τα σημαντικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήσαμε όλοι πως η πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο για να προωθήσει τι συζητήσεις ε, μεταξύ των πολιτών. Πρέπει βεβαίω να είναι κάτι το διάφανο, αλλά και τεχνικά εφικτό από πλευρά Ένωση Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να αναφερθώ μόνο στα επίμαχα τα οποία συζητήθηκαν, δηλαδή η ηλικία ε, των υπογραφών αλλά και το πώς θα προωθήσουμε την ε, συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη. Επίσης ε, για τον έλεγχο του παραδεκτού θα πρέπει να γίνεται πράγματι με την καταγραφή, κάτι το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο είναι το πώς θα αποδειχθεί η εγκυρότητα των υπογραφών μέσω των δεδομένων αυτών. Νομίζω λοιπόν πως το θέμα της ταυτότητας θα πρέπει να εξεταστεί. Ίσως να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος για την ε, ταυτοποίηση. Γιατί νομίζω πως ε, η ουσία είναι το μέσο αυτό να είναι καλό για να προωθήσει την συζήτηση. Οπότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ίσως ε, να μειώσουμε και τον αριθμό των κρατών μελών στο 1 τέταρτο. Κάτι το οποίο επίσης είναι επίμαχο είναι η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά νομίζω πω ο φόβο αυτή τη πλημμυρίδα που αναφέρεται είναι κατανοητός, οπότε εάν επιμείνουμε σε αυτό, νομίζω πάλι πως ο αριθμό των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των καρτών μελών. Αλλά εγώ θα ήμουν κατά του αποκλεισμού των Ευρωβουλευτών από το να είναι μέλη αυτής της Επιτροπής. Αυτό δεν συνεισφέρει στη διαφάνεια και επίσης και οι ευρωβουλευτές, όσο για να σας κάνει εντύπωση, είναι και αυτοί πολίτες. Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι η πρόταση για τον έλεγχο της λεγόμενης πιο ταιριαστή ε, πρόταση, κάτι το οποίο βεβαίω δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσει το αρχικό στάδιο. Και υπάρχει βεβαίω και το θέμα τη αναθεώρηση τη ε, πρωτοβουλία πολιτών. Δεν ξέρω, πέντε χρόνια είναι πολλά, δύο χρόνια είναι λίγα, κάπου στο ενδιάμεσο λοιπόν. Αυτά και σας ευχαριστώ για το εξαιρετικό σα έργο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φοντούν και μετά οι τρεις τελευταίοι ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ γιατί η συζήτηση πραγματικά είναι ιδιαίτερα ζωντανή και το ξέραμε, το ξέραμε ότι θα ήταν έτσι. Γιατί είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Εγώ στην Πολωνία έχω οργανώσει διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό στη δική μου εκλογική περιφέρεια και στη Βαρσοβία πρόσφατα και είναι ένα ζήτημα που πραγματικά προκαλεί συναισθήματα και έντονο ενδιαφέρον. Και ο κόσμος θέλει να ξέρει πότε θα είναι έτοιμη αυτή η δυνατότητα για να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, να συλλέγουν υπογραφές για πολλές ιδέες που είτε θα γίνουν αποδεκτές είτε όχι. Οργανωτική Επιτροπή. Νομικά πρόσωπα. Συμφωνώ θα δούμε βέβαια που θα καταλήξουμε σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα. Εγώ θα προτιμούσα να είναι μεγάλο ο αριθμό, γιατί, Ευρω... γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, άρα θα πρέπει να εκπροσωπούνται και πολλά κράτη-μέλη. Και δεν πρέπει να είναι μόνο άτομα τα οποία είναι ενταγμένα στην κοινωνία τη συγκεκριμένη. Φυσικά πρόσωπα μόνο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα φυσικό πρόσωπο να αρχίζει να σχεδιάζει να συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αν δεν υπάρχει οργάνωση, τέλος πάντων μεταξύ κάποιων φυσικών προσώπων, αν δεν έχουν ε, μια οργάνωση, είναι μια παρέα. Δεν ξέρω ακριβώ τι εννοούσε η συνάδελφο. Θέλετε να υπάρχουν κυβερνητικέ οργανώσει που να είναι μέλη τη Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πρόσωπα τα οποία είναι κατεστημένα ή ίσως είναι και μέλη κάποιας μη κυβερνητική οργάνωσης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει επαφή με πρόσωπα και ευθύνη θα πρέπει να είναι σε άτομα και όχι σε οργανώσει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι, φυσικό, ε, είναι σημαντικό στην Οργανωτική Επιτροπή να συμμετέχουν αυτο λοιπον θεωρω οτι ειναι φυσικο ειναι πρόσωπα. Κάτι είπατε και για βουλευτές. Εγώ δεν μιλούσα μόνο για βουλευτές, μιλούσα για εκλεγμένους πολιτικούς. Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι την πρωτοβουλία αυτή ως ένα εργαλείο για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την νομοθεσία. Και εμείς έχουμε ένα εργαλείο, το κοινοβούλιο, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε στους πολίτες την πρωτοβουλία αυτή. Δεν θα πρέπει να είναι δική μας πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε βουλευτές. Φυσικά και είμαστε και πολίτες, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά νομίζω ότι αν καταλαβαίνω καλά την ιδέα αυτών που συμπεριέλαβαν την πρωτοβουλία των πολιτών στη συνθήκη, νομίζω ότι θέλαν να δώσουν ένα εργαλείο σε αυτούς που δεν είχαν άλλη δυνατότητα να επηρεάσουν την νομοθεσία πέραν της ε, ψήφου τους στις εκλογές. Εμείς είμαστε πολιτικοί, είμαστε εκλεγμένοι και έχουμε και αυτό το μέσο στη διάθεσή μας. Τώρα, να μπουν ε, οι ομάδες άσκησης πίεσης σε αυτό, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα. Ε, το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας ότι μπορεί να υπάρξουν λομπίστες που θα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς τις πρωτοβουλίες αυτής και ίσως να συμβεί αυτό και όταν θα μιλήσουμε για κρατική χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση ή ρύθμιση. Γιατί μια κυβέρνηση, ένα κράτος να δεχθεί όλες αυτές τις ιδέες που θα προκύψουν στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Γιατί θα πρέπει να φέρει την ευθύνη το κράτος λέγοντας ναι αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε, όχι αυτό δεν θα το χρηματοδοτήσουμε. Φοβούμαι ότι δεν θα βρούμε μια ιδεώδη λύση. Όταν μιλώ για χρηματοδότηση, το σημαντικότερο είναι η διαφάνεια. Και δεν μιλάμε μόνο για χρηματοδότηση από εταιρείε, οργανισμούς λοιπά. Είδαμε την εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα και νομίζω ότι η κοινωνία των πολιτών είχε ενεργό συμμετοχή. Με τις ταυτότητες τώρα. Εάν συμφωνήσουμε για την ηλικία από 16 και πάνω. Ότι άτομα δηλαδή ε, από 16 και πάνω μπορούν να υπογράφουν πρωτοβουλίες. Δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν ταυτότητα. Κάποιες φορές έχουν μια σχολική ταυτότητα, παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα τέτοια. Είναι. Και το δεύτερο, δεν χρησιμοποιούν ταυτότητα όλες οι χώρες. Δεν υπάρχει υποχρέωση να έχει κανείς ταυτότητα σε όλες τις χώρες. Άρα δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί την ταυτότητά του να έχει μεν κάποιο έγγραφο αποδεικτικό, κάποιο στοιχείο ταυτοποίηση όταν υπογράφει το να μπορούν να ταυτοποιούν ποιο είναι, αλλά αυτό. Αυτό έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε, ένα ελάχιστο, σε μια ελάχιστη απέτηση. Υπάρχει ένα σύστημα που μπορεί να, να δουλέψει στι ε, τράπεζε, παραδείγματο χάρη. Η ηλεκτρονική υπογραφή δηλαδή. Ε, θα μπορούσαμε όμω να το σκεφτούμε. So, you know, it's not a vote when you talk about the... Μιλάτε για, 16, για τους 16 άριδες. Δεν μιλάμε για ψήφο στις εκλογές. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτοί που υπογράφουν ε, τις πρωτοβουλίες των πολιτών δεν αλλάζουν άμεσα την πραγματικότητα. Ε, δεν είναι το ίδιο με το ότι ψηφίζουν ε, και αν μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, παραδείγματο χάρη. Ουσιαστικά προτείνουν, προτείνουν μια νομοθεσία. Δηλαδή συμμετέχουν άμεσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση, στον ευρωπαϊκό διάλογο. Εγώ θα έδινα αυτή την ευκαιρία στους νέους να μάθουν αυτή την ευθύνη, την ευρωπαϊκή υπευθυνότητα και να δραστηριοποιηθούν. Τώρα, αναθεώρηση. Το σκέφτηκα, για μία μείωση. Νομίζω βάζει την πενταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ προτείνω δύο χρόνια γιατί σκέφτηκα ότι αν βάλουμε δύο χρόνια θα είμαστε ίσως εμεί αυτοί που θα αναθεωρήσουμε. Και θα ήταν ενδιαφέρον εγχείρημα να ξέρουμε αν το έγγραφο το οποίο εκπονήσαμε ήταν καλό ή όχι και αν απέδωσε ή όχι. Βέβαια μέτρησα και τα μήνες και τα χρόνια και τελικά δεν θα είμαστε εμείς. Ακόμα και αν γίνει δεκτή η διετία. Θα είναι μια μακρά διαδικασία. Ίσως η βέλτιστη λύση είναι η τριετία. Και ελπίζω να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Ο ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσουμε και την πρόεδρό μας, την κυρία Ντόρις Πακ. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με αυτό το σημείο όταν ακούσουμε και τους τρεις επόμενους συναδέλφους. Äh, ναι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Φοντούν Βονστάιν για την πρότασή της. Έχω μία παρατήρηση. Ακούστηκε πως είναι σημαντική και η ασφάλεια των δεδομένων. Αυτό αφορά και το διαδίκτυο και τις λίστες. Η διαφάνεια είναι σημαντική, πρέπει να μπορούμε να δούμε ποια δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλίσουμε πως πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το ότι επίσης δεν θα χρησιμοποιηθούν για τίποτα άλλο αυτές οι λίστες, παρά μόνο για την ε, πρωτοβουλία αυτή των πολιτών. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό και στους οργανωτές να μην υπάρχει κατάχρηση. Κάτι άλλο, το οποίο περιέχεται ούτως ή άλλως στο έγγραφο, είναι η διαφάνεια της χρηματοδότησης. Δεν νομίζω όμως πως είναι λογικό να χρηματοδοτεί μόνο το κράτος, αλλά ούτε και μόνο οι οργανώσεις. Σημαντικό είναι να είναι ανοιχτό το ποιος και πώς θα οργανώσει τις πρωτοβουλίες. Αλλά σημαντική είναι η διαφάνεια. Πρέπει να ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί, ποια επιχείρηση, ποιος, ποια οργάνωση, για να μην υπάρχει κατάσταση και από επιχειρήσει και από οργανώσεις. Και τα αναφέρω και τα δύο, γιατί και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν άλλες δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να περάσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό δεν αφορά μόνο τις ε, επιχειρήσεις αλλά και τις ΜΚΟ. Και πρέπει να προσέξουμε όταν θα δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα να αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες έτσι ώστε να αποκλειστούν και επιχειρήσεις και οργανώσεις από την Οργανωτική Επιτροπή. Εάν στηρίζουν επίσης οικονομικά, θα πρέπει να είναι αυτό δυνατό, γιατί από κάπου πρέπει να προέλθουν τα χρήματα, αλλά όπως και δίποτε θα πρέπει να είναι σαφές ότι εμπλέκονται επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε η συγκήτρια να υπάρχει διαφάνεια για να μπορούν και οι πολίτες να αποφασίσουν εάν θέλουν να υποστηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να εμπιστευτούμε τους πολίτες βεβαίως, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα Αυτό είναι... Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι πιστεύω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό φαίνεται και από την συζήτηση που διεξήχθη σήμερα το απόγευμα. Πολλά έχουν δεχθεί, επομένω, δύο παρατηρήσει θα κάνω μόνο. Καταρχά ήθελα να πω ότι εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή, αυτό το άνοιγμα που γίνεται προς τους νέους. Γιατί για μένα αυτό το εργαλείο για το οποίο, το μιλάμε είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αποκτήσει η Ευρώπη και το προσφέρει στους πολίτες της και πιστεύω ότι όλοι οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία που δεν αφορά απλώς και μόνο στις εκλογές, ε, όπως έλεγε και η συνάδελφος, ε, μιλάμε δεν είναι, κάτι, δεν είναι κάτι μελλοντικό που αφορά μια κυβέρνηση, ένα κόμμα κτλ. Είναι, ε, αφορά μια πρόταση που, για θέματα που τους αφορούν άμεσα. Μπορεί να είναι για το σχολείο, μπορεί να είναι για την εκπαίδευση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει ε, τους νέους να τους πάρουμε μαζί μας σε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης ε, για την ε, Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από πολίτες ε, και όχι φυσικά οι νομικά πρόσωπα. Θα μπορούσαμε να βρούμε και μία μέση οδό, δηλαδή να έχουμε μία Οργανωτική Επιτροπή όπου οι πολίτες που θα εκπροσωπούνται εκεί να εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τα θέματα ε, που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της πρωτοβουλία. Δηλαδή να έχουμε φυσικά πρόσωπα και να συνομιλούμε με φυσικά πρόσωπα, αλλά να εκπροσωπούνται και οι οργανώσεις αυτές που ε, θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη ζωή αυτή την ε, ευρωπαϊκής κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την δουλειά την οποία έκανε και για την συζήτηση την οποία προκάλεσε με το κείμενό της. Ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα δημοκρατικό, μια δημοκρατική πρόκληση. Ε, είδαμε ότι στην προεκλογική εκστρατεία και στις εκλογές της ευρωπαϊκές είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό αποχής. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή είναι μια δυνατότητα να έχουμε μια πιο δημοκρατική προσέγγιση. Αρκεί βέβαια να αγγίξουμε όλους τους πολίτες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία για το ψήφισμα πιστεύω το κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο αλλά σαφές. Η σύνταξη δηλαδή να είναι σαφής. Διότι ούτως ή άλλως ε, χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο ε, ε, κοινοτικό και από αυτό το, το λεξιλόγιο θα πρέπει να ξεφύγουμε. Ε, επίσης ψηφιακή επικοινωνία τέλος πάντων. Δεν, ε, είμαστε, δεν είναι όμως όλοι οι πολίτες συνδεδεμένοι με το ίντερνετ, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια επικοινωνία μέσω πολλών μέσων ε, μαζικής επικοινωνίας. Θα πρέπει και οι, οι αγράμματοι και τα άτομα τα οποία δεν έχουν μεγάλη ε, μόρφωση και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Επίσης, ε, για την χρηματοδότηση θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη χρηματοδότηση που γίνεται από, τα, από το κράτος, δηλαδή τη δημόσια χρηματοδότηση, από την συλλογή πόρων μέσω άλλων πηγών. Είναι θέμα διαφάνειας για μένα. Κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπα όλα. Α, επίσης είναι σημαντικό, να έχουμε μια επικοινωνία μαζική. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τι μέσα θα έχουμε στη διάθεσή μας για να φτάσουμε στον πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τούν. Α, όχι. Και κάποιος άλλος ακόμα. Α, ζητώ συγγνώμη. Ξέχασα κάτι ε, που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου ο περιορισμός του αριθμού των κρατών μελών. Εμείς είμαστε υπέρ του ενός τετάρτου και όχι του ενός τρίτου. Η κυρία Φοντούν. Είναι, λοιπόν ζήτημα 7 ή 9 οργανωτών. Εγώ άκουσα από κάποιους πως και 9 είναι λίγοι και πως η πρωτοβουλία πρέπει να εκπροσωπεί την Ευρώπη και όχι λίγα κράτη-μέλη. Φαντάζεστε βέβαια πως κάποιες λίγες μικρές χώρες ε, έχουν ε, κοινά συμφέροντα και θα μπορέσουν να συλλέξουν ένα εκατομμύριο υπογραφές ε, με τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε νομίζω πως όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες επιτροπές θα συζητήσουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Εγώ τίνω προς το 9 Νομίζω πως αυτή η λύση θα ικανοποιήσει και τους περισσότερους. Σύμφωνο πως είναι πάρα πολύ σημαντική η προστασία των δεδομένων. Η Διακομισιόν προτείνει να καταστραφούν αυτές τις υπογραφές μετά από λίγο καιρό. Αλλά αυτό ήταν και ένα ερώτημα που έθεσα και στον εαυτό μου. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα δεδομένα και αν μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Νομίζω πως η μόνη δυνατότητα είναι πως αυτοί που τα συλλέγουν να είναι υπεύθυνοι και όταν φτάσουν τα δεδομένα στην Κομισιόν, η Κομισιόν να τα ελέγξει και να, καταστρέψει να καταστρέψει υπογραφές. Διαφάνεια, μιλήσατε για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι πως οι πηγές πρέπει να είναι ξεκάθαρες και οι πληροφορίες επίσης να είναι διαθέσιμες. Προτείνω λοιπόν να δοθεί η διεύθυνση στο διαδίκτυο, στο έντυπο που θα υπογράφουν οι πολίτες και στη διεύθυνση αυτή να είναι ξεκάθαρη η χρηματοδότηση. Επίσης, φαντάζομαι, προς ε, η πρωτοβουλία αυτή θα χρησιμοποιηθεί κυρίως από ΜΚΟ και όταν μιλάω για φυσικά πρόσωπα, βεβαίως δεν αποκλείει τι δραστηριότητε των ΜΚΟ. Είναι η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά φαντάζομαι κάποιο θα τι υποστηρίζει. Εγώ η ίδια έχω περάσει πολλά χρόνια σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και έτσι είναι τα πράγματα. Είναι η δική μου πρωτοβουλία, την υπογράφω και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μαζί μου που με υποστηρίζουν. Η εκστρατεία πληροφόρηση είναι πρωτοβουλία πολιτών. Ενημερώνουμε τον κόσμο, του πολίτε για το τι κάνουμε, για τα σχέδιά μας κτλ. Όταν μίλησα λοιπόν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως παραδείγματο χάρη την νεολαία σε δράση, τη Europe Direct κτλ. θεωρώ εκεί πέρα πως ε, θα πρέπει να... Εκεί πέρα μιλάμε δηλαδή για την τυπική πλευρά. Τι είναι αυτή η πρωτοβουλία, πώς εκπληρώνονται τα κριτήρια κτλ. Αλλά όταν ξεκινήσει η δράση, μετά επαφίεται στους πολίτες να ενημερώσουν τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων που θα υπογράψουν τα έγγραφα. Και είμαι πεπισμένη πως ε, αυτούς πρέπει να αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο. Το θέμα για τους ανάπηρους και όσους δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ κτλ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σαν την υπογραφή με το διαδίκτυο. που θα συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το λύσουμε τώρα με την πρωτοβουλία των πολιτών, αλλά συμφωνώ πλήρω πω θα πρέπει όλοι να είναι ευαισθητοποιημένοι για το ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα πρόσβασης, ε, ανάγνωσης ή ακρόασης των δεδομένων και να οργανωθούν ε, άρα με τρόπο που θα τους επιτρέπει και σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να λάβουν μέρος. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα το ρυθμίσουμε αυτό με κάποιον τρόπο, αλλά πρέπει όλοι να φροντίσουμε πως η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί. Ε, νομίζω πως απάντησα σε όλα λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τούν. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ όλους όσους απάντησαν. Τώρα θα ήθελα να ακούσω ποιες ιδέες και συναισθήματα προκάλεσε αυτή η συζήτηση στην Κομισιόν. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. <coughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φοντούν για την έκθεσή της, αλλά και όλα τα μέλη για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα αναφέρω κάποια από τα σημεία αυτής της συζήτησης. Καταρχάς, πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την διαφάνεια, για την προστασία των δεδομένων κτλ. συμπεριλαμβάνονται ήδη στην πρόταση της Κομισιόν. Και ήδη τα έχουμε λάβει υπόψη μας για το κείμενο τώρα το οποίο έχει εγκρίνει το Συμβούλιο, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει πάντοτε ένα πρώτο κείμενο το οποίο εγκρίνεται ε, μέσα στα πλαίσια μιας γενικής προσέγγισης, ε, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις της Κομισιόν και τις βελτιώνει. Τώρα, υπάρχει αυτή η ιδέα το, της Επιτροπής των Πολιτών για να εισάγει αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν, ήταν ευρύτερη, πιο φιλελεύθερη, γιατί εμεί θεωρούμε ότι οποιοδήποτε άτομο ελεύθερο, φυσικό, νομικό μπορεί να το κάνει. Η ιδέα όμως την οποία ακούσαμε τώρα ε, τη βρίσκουμε πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα. Ε, για να έχουμε και μια πιο περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση αφενός και για να μην έχουμε και εξωπραγματικές ε, πρωτοβουλίες. Να έχουμε αυτή την Επιτροπή Πολιτών που θα υποστηρίζεται από άτομα βέβαια Βέβαια, καλό θα είναι να ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από την Επιτροπή των Πολιτών, εάν υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει κτλ. Εάν και εφόσον υπάρχουν, ε, για να είναι τα πράγματα τελείω διάφανα. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την δημοσιονομική διαφάνεια, αυτή την εξασφάλισε και η πρόταση της Κομισιό. Ε, η πρόταση τώρα εδώ ε, ενισχύεται, γιατί εμεί είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα αυτά. Πρέπει να θέλουμε να ξέρουμε ποιο πληρώνει. Τώρα για την ηλικία, να σας πω ότι δεν πρόκειται για εκλογές, ούτε καν ένα δημοψήφισμα επίσημο είναι, είναι ε, μια αίτηση προς την, ένα αίτημα προς την Κομισιό να νομοθετήσει σε κάποιον τομέα που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ο χαρακτήρας αυτός του πολίτη ε, και των ε, ε, δικαιωμάτων του πολίτη στην πρωτοβουλία αυτή. Άρα τα κράτη μπορεί να κάνουν αυτό το, αυτή την σύνδεση ανάμεσα στην ηλικία όπου θα επιτρέπεται να υπογράφεται το κείμενο αυτό και την νόμιμη ηλικία. Δηλαδή μπορεί να γίνει και μια παραπομπή στην ηλικία, την νόμιμη ηλικία. Δηλαδή, Οποιοςδήποτε πάνω από 18 μπορεί να υπογράψει, εκτός αν πρόκειται για την Αυστρία, όπου όλοι πάνω από τα 16 μπορούν να υπογράψουν. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω. Τώρα όσον αφορά το αποδεκτό, θα έπρεπε να διευκρινίσω ότι η αρχική μας πρόταση έλεγε ότι αυτός ο έλεγχος αποδεξιμότητας, δηλαδή ο έλεγχος ε, πάνω στη νομική βάση, είναι ο εξή. Υπάρχει η απαραίτητη νομική βάση στη συνθήκη που επιτρέπει την, στην Κομισιό να υποβάλει ε, μια νομοθετική πρόταση. Εκεί μιλάμε για 300.000 υπογραφές. Αλλά το Συμβούλιο τροποποίησε τον αριθμό αυτό και το δεχτήκαμε, αλλά είναι δύσκολο να έχουμε αυτή την διάταξη που διατηρεί το, το ίδιο επίπεδο αξιολόγησης, δηλαδή πραγματική αξιολόγηση της νομικής, της βάσης και ταυτόχρονα να καταργεί α, αυτόν τον αριθμό των υπογραφών, διότι αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο. Καταρχάς η Κομισιό ίσως να είναι υποχρεωμένη καταρχάς να κάνει αυτή την, αυτόν τον έλεγχο, τον εντελεχή έλεγχο και να πάρει μια απόφαση για κάτι το οποίο ενδεχόμενα ποτέ να μην δοκιμαστεί ενώπιον του κοινού, δηλαδή και να μην τύχει καμιά υποστήριξη, ε, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μια ε, δημοσιοποίηση, αν θέλετε, ε, και μια διαφήμιση ότι, η νομοθεσία, ότι δίνεται το πράσινο φως στην Κομισιό μετά, εάν η Κομισιόν ε, καταλήξει στο συμπέρασμα δεν υπάρχει νομική βάση, να φανεί ότι κάνει λογοκρισία. Τέλο πάντων, θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο σα εξηγώ ότι υποβάλαμε την πρότασή μας. Εν συντομία τώρα, επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα, για το ίντερνετ. Το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο στην πρότασή μας, δεν χρειάζεται καν υπογραφή, απλώς συμπληρώνει κάποιος ε, μία αίτηση, ε, δεν, το, δεν την υπογράφει, δεν υπάρχει δηλαδή θέμα ηλεκτρονικής υπογραφής, ε, αυτό ήδη γίνεται και επίσης θέλουμε να έχουμε ένα software, open source software, δηλαδή οι οργανωτές να, έχουν, να οργανώσουν το δικό του site για να συγκεντρώνουν τις υπογραφές. Αυτές, αυτά είναι θέματα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη. Τώρα, τελευταίο θέμα για τις αυτότητες. Δηλαδή, τι έγγραφα θα πρέπει να δείξουν οι υπογράφοντες. Να σας πω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε. Αφορά τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη θα ελέγξουν τα, τις αιτήσει ε, όχι η Κομισιόν και η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών θέλουν να έχουν μια ταυτότητα, ένα αριθμό ταυτότητας. Γι' αυτό και το Συμβούλιο ε, το δέχεται αυτό. Βέβαια το κείμενο του Συμβουλίου είναι έξι σελίδες, το δικό μας κείμενο είναι μονάχα μία σελίδα. Αλλά τέλος πάντων, γιατί εκεί μπήκαν στο, στο σε επίπεδο Συμβουλίου μπήκαν διάφορα, ε, αιτήματα των κρατών μελών τα 21 κράτη-μέλη ε, είπαν ε, ότι θέλουν ταυτότητα και αριθμό ταυτότητα, τα μονάχα τα υπόλοιπα 6 είπαν ότι μπορούμε να ελέγξουμε ταυτότητα των ε, συμμετεχόντων χωρίς την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 1η Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αυτό το σημείο το ολοκληρώσαμε. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, το σημείο Τάκουλα. Ακούσουμε κάποιον που τον ορίζω πολύ καλά από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο και που χαίρομαι ιδιαίτερα που τον ξαναβρίσκω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, τον κύριο Τάκουλα. Να περάσω βέβαια και να αφήσω το, την Προεδρία στην Πρόεδρο, την κυρία Πακ, με την ευκαιρία αυτή. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους μου στην κηδεία του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ο οποίος πέθανε το Σαββατοκύριακο στην ηλικία των 80 ετών και επειδή ήταν φίλος επί 30 έτη καθυστέρησα. Παρακολούθησα λοιπόν την συζήτηση και θεωρώ πως η όλη υπόθεση εδώ πέρα είναι ένα εγχείρημα διαστάσεων που ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν ξέρουμε πώς θα πραγματοποιηθεί και ελπίζω να μην ασχολούμαστε με αυτό όπως ασχολούμαστε με όλα αυτά τα οποία έρχονται στην Ολομέλεια. Εμείς πρέπει να κάνουμε νομοθετικές ε, προτάσεις και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε εκτός. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχει ένας απλός τρόπος να εμπλέξουμε τους πολίτες που δεν θα είναι πολύ πολύπλοκος, αλλά νομίζω πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος βεβαίως μέχρι να έχουμε μια σωστή πρόταση. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά. Χάνου Τάκουλα, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι είμαστε λίγο πίσω στο χρόνο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συντομεύσω την παρουσίασή μου. Εδώ μιλούμε για την ένταξη των Ρωμά στο κοινωνικό επίπεδο. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση, την οποία θα αναλάβει η Επιτροπή Ελευθεριών. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με, με τα διακοσμητικά στοιχεία, αλλά με την ουσία, με αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί στην στάση μας εδώ. γιατί πραγματικά τις τελευταίες εβδομάδες είδα ότι δεν υπήρξε και ιδιαίτερη σοβαρότητα στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι υπερψήφισαν, κάποιοι καταψήφισαν ε, τη συμπεριφορά της γαλλικής ε, κυβέρνησης. Και ίσως και κάποια μέτρα που ακόμη και αν δεν κοστίζουν υπέρ των Ρώμα δεν τα υπερψήφισαν. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή μας είναι μια πολιτισμένη Επιτροπή παρόλα αυτά. Και αν λέμε κάτι πρέπει και να το λέμε αλλά και να το κάνουμε πράξη, να το μετατρέπουμε τα λόγια σε έργα σε επίπεδο των κρατών μελών. Αυτό είναι το ουσιώδες. Πρέπει να κάνουμε πράγματα υπέρ της κοινότητας των Ρωμά. Τον τελευταίο καιρό, όπως και φαντάζομαι υπόλοιποι συνάδελφοι, ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο αυτό θέμα και είδα ότι υπήρχαν σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα. Εκπαίδευση. Γνωρίζω ότι είμαστε 27 κράτη-μέλη, άρα έχουμε 27 διαφορετικές στρατηγικές υπέρ της εκπαίδευσης των Ρωμά. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να εξετάσουμε κάποιες πρακτικές, να δοκιμάσουμε κάποιες καλές πρακτικές σε επίπεδο εκπαίδευσης, για να αποφύγουμε τη διακριτική μεταχείριση και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αναπτύξουμε και μια στρατηγική. Σας θυμίζω ότι είναι πολύ η κοινότητα των Ρώμα. Είχαμε κάποιες ε, αποτυχίες μέχρι τώρα. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ άριθμη, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κοινότητα αυτή με ελαφρότητα. Η Επιτροπή Ελευθεριών θα δει και τα δικά της δήματα και εμείς θα δούμε τα σχετικά με την νεολαία, την παιδεία, τον πολιτισμό, θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Φαντάζομαι ότι κομβικό σημείο είναι η εκπαίδευση και από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Κάτι άλλο που δεν θα πρέπει να ξεχνούμε είναι και η δύναμη ε, της ένταξης μέσω του αθλητισμού. Είναι μια πρακτική που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται και γιατί όχι για τους μετανάστες ε, και γιατί όχι και για τους Ρωμά. Αν λοιπόν εγώ έπρεπε να επιμείνω σε κάτι, θα επέμενα στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνουν συζητήσεις και ελπίζω να είναι εστιασμένες και στοχευμένες αυτές οι συζητήσεις. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να ξέρω είναι ποια είναι τα ουσιαστικά τα βασικά σημεία που θα πρέπει να συμπεριλάβω στην έκθεση, να συμπεριλάβουμε στην έκθεση μας στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι μου δημιουργεί ντροπή ε, όταν βλέπω αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη, γιατί πολλές φορές δίνουμε μαθήματα από εδώ και από εκεί, αλλά από την άλλη κάποιες φορές ε, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση που επιφυλάσσουμε εμείς ορισμένες μειονότητες, ε, κάποιοι άλλοι μας δείχνουν το δάχτυλο. Δίνουμε και στους Παλαιστινίους κάποια μαθήματα και επίσης δίνουμε και ε, χρήματα, δεν δίνουμε όμως πολλά για την ένταξη των Ρωμά. Θα πρέπει να διορθωθούν όλες αυτές οι αδυναμίες και ανεπάρκειες, αλλά κατά την άποψή μου θα πρέπει να παραμείνουμε στα πιο ουσιώδη για την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. πως έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα συχνά στην Επιτροπή μας ε, και ο κ. Στάκουλα έχει γράψει και μια έκθεση για την ένταξη των μεταναστών. Οπότε νομίζω πως είστε ο σωστός συντάξης γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Βέβαιω είναι εκρηκτικό αυτή τη στιγμή γιατί εγκρίναμε και το ψήφισμα για τις απελάσεις από την Τώρα, Herr Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό αλλά και λεπτό το ζήτημα αυτό και είναι πολύ εύκολο κανείς ε, να ε, είναι δημαγωγός ίσως ε, και λαϊκιστής με αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που πρέπει κυρίως να μιλήσουμε είναι για τη βούληση ενσωμάτωσης και ένταξης. Για τη βούληση των ίδιων των μελών της κοινότητας αυτής να μορφωθούν, να εκπαιδευτούν. Έχουμε εμείς μια σημαντική κοινότητα τσιγκάνων ε, στην Ισπανία, που ουσιαστικά είναι ενταγμένη ε, στη χώρα, σχεδόν ε, θα έλεγα πλήρως ενταγμένη στην Ισπανική κοινωνία. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο με τους Ρωμά. Και με τη συνάδελφό μου, την Μαρία Τερέσα, Επισκεφθήκαμε την ε, Μπανταλώνα στα περίχωρα της Βαρκελόνης ε, με 120.000 κατοίκους πρόσφατα. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Ρωμά που δεν ζουν σε καταβλισμό αλλά σε σπίτια ε, με τον τοπικό πληθυσμό δηλαδή ουσιαστικά επιβιώνουν αλλά υπάρχουν προβλήματα, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής αυτής και όταν μιλά κανείς με αυτού βλέπει πόσο δύσκολη είναι η ε, οποιαδήποτε αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευσης, δεν είναι ότι δεν θέλει ε, η κοινωνία να κάνει κάτι για ε, αυτή την κοινότητα, είναι ότι οι Ρωμά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ενταχθούν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και σημαντική προσπάθεια στις χώρες ε, καταγωγής των Ρωμά, οι οποίοι λαμβάνουν πολύ σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν τα χρησιμοποιούν για την ένταξη ακριβώς των Ρωμά στις χώρες καταγωγής τους. Ίσως αυτό που λέω να ακουστεί σκληρό και δύσκολο να το δεχθούμε. Αν θέλουμε όμως να το εκμεταλλευτούν τα ακροδεξιά κόμματα και ξέρουμε ότι πολλοί πολίτες μας ψηφίζουν αυτά τα κόμματα. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να το εκμεταλλευτούν θα πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Θα πρέπει να δείξουμε σθένος, αποφασιστικότητα όταν συζητούμε για το θέμα αυτό. Πράγματι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το ζήτημα αυτό και πολλές φορές προκαλεί αντιπαραθέσεις όταν μιλάμε πλέον για διακρίσεις. Πάντοτε νομίζω ότι όπως το προσεγγίζουμε το ζήτημα, κάποιες φορές στιγματίζουμε από μόνιμους πληθυσμούς ε, για τους οποίους, ε, στους οποίους αναφερόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να προσέξει ο πού απευθύνεται ακριβώς. Εμείς είμαστε Επιτροπή Πολιτισμού. Το πρώτο πράγμα πρέπει ε, να ξέρουμε για ποιο πληθυσμό μιλάμε. Πώς ορίζουν οι ίδιοι οι Ρωμά. τον εαυτό τους. Εμένα ο ορισμός των Ρωμά ε, στα διάφορα διεθνή φόρα μου αρκεί και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε θετικά και να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον πληθυσμό. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά όλες τις πολιτιστικές μειονότητες, εάν Πρώτα και πάνω από όλα αυτό που θέλουμε είναι να επιβάλλουμε το δικό μας μοντέλο και δεν σεβόμαστε την πολιτισμική διαφορά και διαφορετικότητα, δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα πάμε πουθενά. Για να προχωρήσουμε πρέπει να αναγνωρίζουμε τον πλησίον μας, να αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητά του και να πάψουμε να προβαίνουμε σε διακριτική μεταχείριση όταν ο άλλος δεν μοιάζει με εμά. Είναι νομίζω το α και το ω. Και ένα τελευταίο στοιχείο για το οποίο θέλω να, στο οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξή. Δεν αρκεί να δίνει πόρους, να δίνει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι αποτελεσματική και η αντίστοιχη πολιτική της. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό ε, είναι ε, αντίθετα και το παράδειγμα προς αποφυγή θα έλεγα. Γιατί όπως λένε και οι αρμόδιοι επίτροποι, τα χρήματα τα οποία προορίζονται για τους Ρωμά τελικά δεν αξιοποιούνται. Και η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι γιατί. Γιατί δεν αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα. Μήπως οι κυβερνήσεις που τελικά είναι ε, από τις οποίες προέρχονται βασικά η ε, διακριτική αυτή μεταχείριση. Και δεν θέλω να φέρω συγκεκριμένα κράτη. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτά τα κράτη, τα οποία ε, δεν ε, φέρονται αντικειμενικά, ας πούμε, έχουν μια διακριτική μεταχείριση, μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ο Μάρκο, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έρχεται στο σωστό χώρο η έκθεση αυτή και είναι και πολύ επίκαιρη δεδομένη όλες όλη συζήτηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν θα πρέπει να είμαστε δογματικοί και θα πρέπει να μιλήσουμε για τα ζητήματα τα οποία εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, πολιτισμός αλλά και κυρίως εκπαίδευση όπως είπε ο εισηγητής και αθλητισμός όμως, ναι είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά φυσικά και στο θέμα αυτό θα πρέπει να συμφωνούμε. Η σχολική εκπαίδευση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες τοπικές αυτοδικήσεις οι οποίες δαπανούν τεράστια κονδύλια ε, για την εκπαίδευση των Ρωμά, αλλά δυστυχώς παραμένουν κενά τα έδρανα που απευθύνονται, που προορίζονται για τους Ρωμά. Διότι οι οικογένειε αυτέ αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Δεν λέω ότι τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, αλλά οι οικογένειε αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και δεν πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά του. Το σχολείο όμω είναι ουσιώδε, είναι ίσω το πρώτο βήμα. Αν θέλουμε λοιπόν να ενταχθούν τα παιδιά αυτά, πρέπει να πάνε σχολείο. Αλλιώ ούτε δουλειά θα βρουν, ούτε ρόλο στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Έχω δει πολλά σχολεία όπου τα παιδιά περνούσαν από τη μια τάξη στην άλλη χωρίς να καταλαβαίνουν καν τη γλώσσα στην οποία γινόταν η διδασκαλία και χωρίς να έχουν αφομοιώσει καθόλου τη διδακτέα ύλη προηγούμενης χρονιάς. Αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος βέβαια. Τα άτομα αυτά σίγουρα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμά τους, ταυτόχρονα όμως να φροντίσουμε να ενταχθούν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Αλλιώς λέμε λόγια του αέρα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ανταλλαγή ιδεών, απόψεων για την εκπαίδευση, για τα σχολεία. Και να αφήσουμε κατά μέρο τα δόγματα και τι ιδεολογίε. Να προσπαθήσουμε να υπάρχει πραγματική ενσωμάτωση, πραγματική ένταξη. Ευχαριστώ. Tämä on asia ja nyt kun Ευχαριστώ. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο αυτό το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση βιάστηκε πάρα πολύ. Θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες τις ε, προενταξιακές. Π.χ. η Σλοβακία υπήρχαν τέτοιες, τέτοια προβλήματα πριν από λίγα χρόνια, αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τόσο δύσκολη που δεν πρέπει να βάζουμε ετικέτες σε μια ομάδα ανθρώπων. Γιατί αν σκεφτούμε οποιοδήποτε πληθυσμό, υπάρχουν πάντα αυτοί που τα πάνε καλύτερα από τους άλλους, κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Ο κύριος Στάκουλα ξέρει τι γίνεται στη Φιλανδία, πολλοί Ρωμά είναι μια χαρά ενταγμένοι στην κοινωνία, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς εγκληματίες. Οπότε δεν μπορούμε όλους μαζί να τους βάλουμε σε ένα τσουβάλι και είναι και θέμα κυριαρχίας. Έχουν οι χώρες το δικαίωμα να αποφασίσουν ε, ποιον δέχονται στην επικράτειά τους και ποιον όχι. Και από την άλλη πρέπει να δούμε και το θέμα της ελευθερής διακίνησης. Οπότε πρέπει να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα σε αυτά. Κύριε Κώστα. Ehm, mm, Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή και έρχεται και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Διότι διακυβεύονται εδώ θεμελιώδεις αξίες και αρχές. Η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να συμβάλλει κατά τρόπο που να εμβαθύνουμε στα πράγματα. Αλλιώς να πούμε απλά ότι η ένταξη δεν είναι δυνατή. Η ευθύνη μας είναι αυτή. Φυσικά και δεν νομίζω, κύριε Τάκουλα, ότι θα καταλήξουμε στη δεύτερη επιλογή, να πούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης. Πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε σε μια συζήτηση που γίνεται σε ένα ιδιαίτερα δραματικό πλαίσιο, θα έλεγα, ε, και με τόσα προβλήματα ένταξης. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε η Επιτροπή Πολιτισμού. Επομένως, πρέπει όπως και δίποτε να εγκύψουμε στη διαπολιτισμική πτυχή του θέματος. Πρέπει να εμείνουμε στις ιδέες και στις αξίες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Προσωπικά δικαιώματα, μη διακριτική μεταχείριση και σεβασμό των μειονοτήτων, αυτό είναι ουσιώδες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι πάντοτε σεβόμενοι το δίκαιο κτλ. Θα πρέπει να προασπίζουμε, να υπερασπίζουμε και το δικαίωμα της ένταξης των πληθυσμών αυτών. Δεν συμφωνώ όταν ακούω ότι η ίδια η κοινότητα των Ρωμά ε, έχει κάποιες επιφυλάξεις και δισταγμούς απέναντι στην ένταξή της. Αν μιλάμε για ένταξη πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις ε, εκ των ουκάνευ προϋποθέσεις. Και όταν μιλάμε για Ρωμά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις διαφορές, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και πρέπει να πω ότι σήμερα και μιλάμε και για την δυνατότητα μετακίνησης και την ελευθερία μετακίνησης των Ρωμά στην Ευρώπη, εφόσον πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή λοιπόν η έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει να αναφέρει και κάποιες θετικές εμπειρίες ένταξης από ορισμένε χώρες. Ο κύριος ε, Σοήνη έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν πρέπει να ε, δείχνουμε με το δάχτυλο την τάδε ή τη δίνα χώρα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να, κάνουμε, να βρούμε κάποια στοιχεία κοινά μεταξύ ορισμένων κοινοτήτων και των Ρωμά, όπως το χάρη αστικών ε, περιφερειών. Στην, ε, στο Τρεντίνο, παραδείγματο χάρη, έκλεισαν κάποιοι καταβλισμοί και οι Ρωμά ε, εκπαιδεύτηκαν και τα λοιπά και τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά. Δεν είναι βέβαια η μόνη δυνατότητα, αλλά υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα, κάποιες θετικές εμπειρίες. γιατί ή θα δημιουργήσουμε τελικά ένα πρόβλημα δημόσιας τάξης που θα ήταν λάθος, ή θα πούμε το αφήνουμε κατά μέρο, δεν μπορούμε αυτό το θέμα να το θίξουμε. Όχι, ούτε η μία οδό είναι σωστή, ούτε η άλλη. Πρέπει να βρούμε την τρίτη οδό, να βρούμε μέσα και τρόπους να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φαντάκουλα, βεβαίω. Δεν θέλω να προσθέσω μόνο μία σκέψη. Υπόθηκε πω. Ε, ναι, ο Χάνου πρέπει να φύγει πως δεν είναι ευχάριστα τα οράματα και δεν ξέρουμε με την εφαρμογή. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε εκεί όπου ζουν οι Ρώμα, να δούμε πώς θα έρθει ο πληθυσμός αυτό σε επαφή με τους Ρώμα και να αναλάβουν, ξέρω εγώ, ένα παιδί για να το πάνε στο σχολείο. Και αν πηγαίνει κάποιος τρεις μήνες με ένα παιδί στο σχολείο, θα βλέπει πως μπορεί να μάθει κάποια πράγματα, θα φροντίζει να ανατρέφεται σωστά, να δημιουργηθούν δηλαδή έτσι δυνατότητες επαφή των ανθρώπων στο τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει σε κάποιους δήμους, αλλά υπάρχουν και κάποια υποδείγματα και έτσι, παραδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, αν, αν είστε γρήγοροι, σας παρακαλώ, ε, μπορείτε να μιλήσετε γρήγορα γιατί πρέπει να φύγει ο Χάνο Τάκουλα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι όπως ε, πρέπει να χειριζόμαστε τον όρο Ρωμά με προσοχή, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τη λέξη διακριτική μεταχείριση. Φυσικά και θα πρέπει να σεβαστούμε την πολιτιστική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει σήμερα ένα πρόβλημα με το μοντέλο των Ρωμά, αφού έτσι πρέπει να τους λέμε, και αν έχουν δυσκολίες αφομοίωσης και ένταξης, μάλλον ένταξης, σας παρακαλώ κυρία μου, εγώ σας άκουσα. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται έχουμε ένα πρόβλημα σεβασμού, αμφίδρομο και προς τις δύο πλευρές, ε, όχι μόνο προς την πλευρά των Ρωμαίων. Εσείς δεν σέβεστε αυτόν που μιλάει πάντως σίγουρα, κυρία μου. Λοιπόν, Έχουμε τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά η ε, κυρία Κώστα λέει ότι ε, ίσως ε, για κάποιους ε, είναι αδύνατη η ένταξη και νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις στέφθηκε με αποτυχία η προσπάθεια ένταξης. Σίγουρα μέσω της παιδείας και της και του πολιτισμού μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή πρακτικών, να εμπνευστούμε από αυτά που έχουν εφαρμοστεί και λειτουργήσαν. Σίγουρα να καταδικάσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα και να πω ότι αυτό που συνέβη στη Γαλλία ε, σας ζητώ να μην το κρίνετε γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό, αλλά σίγουρα πρέπει να ε, θίξουμε τα πραγματικά προβλήματα και να αναλάβουμε δράση. Πρόεδρος, ναι πράγματι, Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων και όχι για να κατηγορούμε τους πάντες. Χάνου τάκουλα. Τελευταία σου λέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για το ότι θα πρέπει να φύγω σύντομα. Κέταξα το πρόγραμμα. Ε, θα επιστρέψω. Κοιτάξτε, νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Χρειαζόμαστε τώρα ένα πιλωτικό, αν θέλετε, έργο, σχέδιο και έχω καταθέσει και μία πρόταση για τον προπολογισμό για να μπορέσουμε να βρούμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Αλλά αν μόνο μιλάμε για αυτά τα πράγματα και ακόμα κι εσείς ε, είπατε πως είστε κατά, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Στην Ανδία τα έχουμε πάει σχετικά καλά με την ένταξη. Εγώ σπούδασα στη Φιλανδία και είχα πολλούς συμφοιτητές Ρωμά. Οπότε δεν θεωρώ πως είμαστε και καμία εξαίρεση στον τομέα αυτόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν το ευρωπαϊκό μοντέλο βλέπετε εδώ πέρα και μέσα συζήτηση εδώ μέσα υπάρχουν εντάσεις. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δράση οπωσδήποτε. Οπότε θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλα όσα ακούστηκαν και να πούμε πως ε, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για να έχουν δυνατότητα μια καλή ζωή τα παιδιά των Ρωμά, να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τέλος να πω πως αυτό είναι σημαντικό γιατί ε, εμείς οικοδομήσαμε την Ευρώπη στις τάχτες του ολοκαυτώματος. Ε, 6 εκατομμύρια Εβραίοι και 500-600 χιλιάδες Ρωμά δολοφονήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει η πρόεδρος. Έχουμε ακόμα την κυρία Μπενέρα αυτού, η οποία θέλει να γράφει το λόγο. Je voudrais simplement insister sur une chose. Nous sommes dans la, euh, dans la commission culture et nous n'avons pas parlé de la culture rome. Moi, je voudrais insister là-dessus.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 Moi, je pense que si on veut qu'ils viennent vers nous, il faut qu'on va vers eux. Et ça, on n'a pas parlé de ça. Et je pense que c'est dommage, parce que les Roms ont une culture très forte. Liebe Frau Benarabtou, daran zweifeln wir nicht. δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην κοινωνία μας τους Ρώμα. Δεν μπορούν να είναι μια χωριστή κοινωνία, πρέπει να ενσωματωθούν. Δεν χάνουν έτσι τον πολιτισμό τους. Προσπαθούμε να υιοθετήσουμε τα απαραίτητα σε μια χώρα στην οποία πρέπει να δεχτεί κανείς αν ζει σε μια χώρα. Π.χ. πρέπει να πάει στο σχολείο. Όταν λέει ο κύριο Στάκουλα να πηγαίνουμε τα παιδιά σχολείο, αλλά θαυμάσιο, αλλά εγώ ξέρω. Ε, υπάρχει μια γειτονιά μου, στη γειτονιά μου, ένα καταβλισμός Ρώμα, τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο. Πρέπει δηλαδή να βρεθούν κάποιοι νονοί, αν θέλετε, αυτών των παιδιών, που θα τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν. Αυτό χρειαζόμαστε. Οπότε χρειάζεται βοήθεια και συμπόνια για αυτούς τους ανθρώπους και όλες οι ενώσεις, όλες οι οργανώσεις που υπάρχουν επί τόπου να μπορέσουν να βοηθήσουν έτσι ώστε να βρουν οι άνθρωποι αυτοί το δρόμο τους προς την κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως χάνουμε την ταυτότητά τους, κάθε άλλο. Μπορούν να την εκφράσουν καλύτερα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο λοιπόν. Λοιπόν, ε, κύριε Καβαντά, ορίστε να μιλήσουν όλοι οι Γάλλοι. Μιλήστε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ζητήσει και από πριν το λόγο. Αλλά ίσως να μην, ήμουν, να μην κουνήθηκε αρκετά και να μην με είδατε. Την άλλη φορά θα το κάνω καλύτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξω κάποια θέματα για μια ε, συζήτηση που έγινε κάτω από ήρεμους τόνους. Η Ρωμά είναι ενδο, και είναι καθαρά ευρωπαϊκός λαός. Τώρα, θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα αυτούς που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μια χώρα και αυτούς που θέλουν να παραμείνουν νομάδες δηλαδή να μεταναστεύουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν δύο, δύο περιπτώσεις, δύο καταστάσεις. Είναι η συνηθισμένη κατάσταση σε, που ισχύει σε πολλέ χώρε στην Ισπανία, στην Αυστρία, όπου οι Ρωμά οργανώθηκαν και έχουν εκπροσώπους, έχουν ενώσεις με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή εκεί η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να τους εντάξει, επομένως η ένταξη λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Στην Ισπανία είναι η καλύτερη, ε, το καλύτερο παράδειγμα. Εκεί έχουμε μια αστική τάξη Ρωμά δικηγόροι, γιατροί κτλ. Όχι μόνο μουσική, έστω και αν είναι ένα μεγάλο μέρος του, της κουλτούρας τους η μουσική. Και μετά υπάρχει και η άλλη πτυχή, που είναι η φτώχεια. Για τους ε, μόνιμα εγκατεστημένους Ρωμά. Είναι κρατικό το θέμα με την ε, βοήθεια των Ευρωπαϊ... της ευρωπαϊκής ε, κοινότητας, τη χρηματοδότηση που δίνει η Ευρώπη. Πολλές φορές η χρηματοδότηση αυτή δεν φτάνει ποτέ στους Ρωμά. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπάνω. Και σε αυτή την θητεία και στην προηγούμενη, το θίγουμε το θέμα. Στην προηγούμενη ε, θητεία, όταν ήμουν ε, πρόεδρος της Επιτροπής Λιμπέ, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε κοινωνικά, κοινοτικά κείμενα για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και η εκτελεστική εξουσία της κοινότητας και κάποιες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου μας σταμάτησαν. Η κυρία Βικτόρια Άτσε που ήταν ε, ε, βουλευτής Άλντε στην προηγούμενη θητεία ήθελε να φτάσουμε κάπου και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε διότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα καθεστώς Ευρωπαίων μετακινούμενων. Δηλαδή είναι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι απόλυτα νόμιμοι, ε, αλλά που δεν θέλουν να κατασταθούν σε ένα κράτος, αλλά θέλουν να, μετακινούν, μετακινούνται. Δηλαδή για τους μόνιμα εγκατεστημένους υπάρχουν τα, υπάρχει μια ρύθμιση, υπάρχει μια πρόβλεψη. Για τους μετακινούμενους τι, τι υποχρεώσεις, τι δικαιώματα έχουν θα πρέπει να έχουν τα δικαιώματα που, έχουν κάθε, που έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης με ένα διαβατήριο μετακινούμενου. Τώρα οι υποχρεώσεις τους ποιες είναι. Θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει υποχρέωση εκπαίδευσης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό μέσω των οργανώσεων Ρωμά. Ποια, ποιος είναι ο πολιτισμός, ποια είναι η κουλτούρα που πρέπει να πάρουν τα παιδιά αυτοί και θα πρέπει να ξέρουμε για ποια είναι τα υποχρεώσει και τα δικαιώματά του ε, σαν Ευρωπαίοι πολίτε. Μετά, ένα άλλο θέμα είναι η υγεία. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα υγειονομική περίθαλψης. Και άλλο ένα σημείο είναι η ασφάλεια. Θα πρέπει να σέβονται τους όρους και την ε, ασφάλεια μιας χώρας όπου είναι κατεστημένοι, ε, που βρίσκονται και από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη δική τους ασφάλεια γιατί σε κάποιες χώρες γύρω από τον Δούναβη, εκείνοι αποτελούν ε, θύματα επιθέσεων. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι πολύ σοβαρό, κυρία Πρόεδρε, και είναι καθαρά ευρωπαϊκό θέμα. Φύσας, τελευταία λέξη. Να κάνω μία σύντομη παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Καβαντά. Αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην Ισπανία είναι οι Ισπανοί τσιγκάνοι. Έχω φίλους τσιγκάνους που ασχολούνται με την μουσική ή που είναι γιατροί ή δικηγόροι. Αυτοί είναι απόλυτα ενταγμένοι στην ισπανική κοινωνία. Οι δυσκολίες όμως που έχουμε δεν είναι με αυτούς τους τσιγκάνους, είναι με τους Ρωμά. Και Ρωμά α, εμείς ονομάζουμε αυτούς που έρχονται από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, Βουλγαρία και Ρουμανία και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ενταχθούν. Δηλαδή υπάρχουν και προβλήματα ανάμεσα στους Ισπανούς τσιγκάνους και αυτούς που έρχονται από, από το εξωτερικό. Γιατί και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι καλές. Εμείς στη Γερμανία έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για Ρώμα δεν ε, μπορούμε να του λέμε τσιγκάνους, ε, οπότε μιλάμε μόνο για Ρώμα ε. και Σύντη και μάλλον για Ρώμα μόνο. Και εκεί υπάρχει άλλη μια ομάδα που έχει άλλο όνομα, που έχει ίσως και διαφορετική ιστορία, ανήκει τέλος πάντων στη μεγάλη ομάδα των τσιγκάνων όπως λέγαμε παλιά, δεν, το λέω τώρα έτσι με την κακή έννοια, οπότε μιλάμε και για τσιγκάνικη μουσική, εν πάση περιπτώσει κάποιοι τσιγκάνοι θα παίζουν και αυτή τη μουσική. Λοιπόν, όπως είπαμε είναι πολύ επέδο και δύσκολο το πρόβλημα. Ο κύριος Στάκουλα σωστά τα είπε και πράγματι καλό θα ήταν να συνεννοηθεί και με τον κύριο Καβαντά για το πώς θα μπορέσει η έκθεση να συμπεριλάβει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπαν οι Γάλλοι συνάδελφοι. Αυτά σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα άλλο. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πρόταση του κύριου Σκουρίγια για... και κατόπιν αυτής της πρότασης ε, προσκαλέσαμε τον κύριο Τζιάν Φραντσέσκο Λιπατέλη, Προέδρου της ΑΣΕΣ Europe και όπως ξέρετε το θέμα είναι ο αθλητισμός ε, που υπάρχει πλέον στη συνθήκη με την Λισαβόνα, αλλά δεν θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα με το πρόγραμμα εδώ του αθλητισμού, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και δεν έχει και πολύ διάθεση το Συμβούλιο. Αλλά θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Ίσως μπορούμε σήμερα, δεν ξέρω, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τι θα κάνει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε τον κύριο Λουπατέλη. Το όνομα του δεύτερου κυρίου δεν το ξέρω. Πρέπει να συστηθείτε. Έχετε από 15 λεπτά, όχι έχετε 15 λεπτά και οι δύο για να κάνετε μια εισαγωγή στο θέμα σας και μετά θα έχουμε άλλα 15 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριε Λουπατέλη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε αυτό την Ευρωπαϊκή Οργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σίλβια Κώστο, τον, τον Μάρκο Σκουρίγια και άλλους φίλους βουλευτές που αγαπούν τον αθλητισμό ε, και τους πολίτες. Αυτή η πρωτοβουλία που αναλάβαμε, Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες ε, για τον, ε, για τον Αθλητισμό, είναι μια δέσμευση που, ανα, που αναλάβαμε να προωθήσουμε τον αθλητισμό σε όλες τις χώρες γιατί είναι, για να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ευσοία των, των πολιτών. Ευχαριστούμε την κυρία ΠΑΚ για την πρόσκληση αυτή. Είναι εδώ μαζί μας και εκπρόσωποι της, ε, της ε, Ισταμπούλ, της, του Κάρντιφ και Αμβέρσας, που είναι οι, οι τρεις ε, πόλεις υποψήφιες για την, για την πρωτεύουσα, αθλητική πρωτεύουσα του 2012. Ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία αυτό το 1999 στη Μαδρίτη και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε μια, να ε, ενωθούμε μια ομάδα αθλητικών ομοσπονδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, να δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Αθλητισμού. Το ξεκινήσαμε στη Μαδρίτη με τον ε, Αλβάρες Δεμανσάνο που τότε ήταν δήμαρχος της Μαδρίτης και που ήταν ιδιαίτερα δεσμευμένος ε, με τον αθλητισμό. Πάνω από 300.000 μαδριλένοι ε, ε, χρησιμοποιούσαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαδρίτης, τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάναμε μία ανάλυση ευρωπαϊκό επίπεδο και το 2001 η Μαδρίτη αποτέλεσε την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του αθλητισμού. Το να είναι, κανείς, ε, το να είναι μια πόλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του αθλητισμού σημαίνει πολλές δεσμεύσεις, διότι οι πόλεις ε, αυτές από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου θα πρέπει να οργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες για τους πολίτες τους. Αυτά τα 11 χρόνια προχωρήσαμε τις δεσμεύσεις, τις μας και μετά την Μαδρίτη από το 2001 είχαμε τη Στοκχόλμη, Γλασκόβη, Αλικάντε, Ρότερνταμ, Στουτγκάρδη, Κοπενχάγη το 2007, ε, Στουτγκάρδη, ε, Βαρσοβία, Μιλάνο, Δουβλίνο και η δέσμευσή μας είναι να ε, βοηθήσουμε τους πολίτες μας να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό για το καλό το δικό τους, αλλά και για το καλό όλων και για το γενικότερο καλό. Και δίνω τον λόγο τώρα στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λουπατέλη. Θα σας περιγράψω λίγο περισσότερο τις δραστηριότητες. Όπως είπε και ο Πρόεδρος Λουπατέλη, η βασική ε, η δραστηριότητα είναι να αναθέσουμε, την, να αναδείξουμε την πρωτεύουσα του αθλητισμού, το βραβείο αυτό αν θέλετε, αλλά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες Η δεύτερη βασική δραστηριότητα μας είναι ότι εδώ και λίγα χρόνια η Ένωση έχει ε, συντάξει, έχει αποφασίσει αυτό το πιστοποιητικό ποιότητας για αυτούς που ασχολούνται με τον ε, και διδάσκουν τον αθλητισμό Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουμε, όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις, στους Δήμους και τις κοινότητες, η προετοιμασία ενός παρατηρητηρίου για τις πρακτικές του αθλητισμού σε επίπεδο τοπικό. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι μία από τις βασικές ε, βασικά χαρακτηριστικά μας είναι ότι κάνουμε μια συνολική εκτίμηση όταν αποφασίζουμε ποια θα είναι η πρωτεύουσα του αθλητισμού. Κάθε χρόνο μία εκλέγεται. Είδαμε το 2011 ήταν η Βαλένθια. Η... Τέλος Νοεμβρίου θα αποφασίσουμε ποια θα είναι η πρωτεύουσα του 2012 και έχουμε εννέα πόλεις ε, κάθε χρόνο που παίρνουν κάποιο βραβείο. Ε, και μικρότερες πόλεις, δεν έχουμε μόνο τις πρωτεύουσε. έχουμε και 100.000 πόλεις, μικρές ή μικρότερες, ε, μη μεγαλύτερες, που ε, μπορούν να ε, επιλεγούν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Αθλητισμού. Εδώ έχουμε συμπεριλάβει μία σύνοψη της διαδικασίας επιλογής ε, είναι, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Μπορείτε να μπείτε στο site μας και να δείτε ακριβώς τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία κρατάει πολλού πολλούς μήνες και που επιτρέπει σε όλες τις πόλεις, μικρές και μεγάλες, να πάρουν το βραβείο αυτό. Ε, αν θέλετε μπορούμε να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μια άλλη δραστηριότητα είναι αυτή την οποία ανέφερα προηγουμένως, που είναι το πρόγραμμα για ένα πιστοποιητικό ποιότητας ε, των ε, αθλητικών ε, διευθυντών, αν θέλετε, σε επίπεδο τοπικό. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά το θέμα, τα θέματα διαχείρισης του αθλητισμού σε επίπεδο πόλης. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται παράλληλα με την ε, ανάδειξη της ε, πρωτεύουσας και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τώρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ε, ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις πόλεις, πρακτικών που αφορούν την ε, την διαχείριση του αθλητισμού. Έχει υπογραφεί μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της Πίζας και της Μαδρίτης ε, για να γίνει μια πιο λεπτομερής μελέτη του θέματος και ε, τα επόμενα χρόνια θα είναι, πιο, θα είναι καλύτερο αυτό το πιστοποιητικό. Τώρα, ξέρετε όλοι ότι το ASES είναι μια πρωτοβουλία ε, η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα σαν ε, πεντηκοστή δράση στην Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό. Και ξέρετε ποια είναι τα ποσοστά των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και εντός και εκτός αθλητικών ομίλων. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να, να ολοκληρώσουμε μια προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού και χάρη στα δίκτυα τα οποία έχουμε, 70 ε, πόλεις έχουν συμμετάσχει στο δίκτυο, ε, χάρη στο δίκτυο αυτό, το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος του Πατέλη, θέλουμε να προωθήσουμε τον εθελοντισμό στον αθλητισμό συνειδητοποιήσαμε και εδώ πρόκειται για ευρωπαϊκές εκθέσεις ε, που το τόνισαν αυτό ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον εθελοντισμό στις, ε, ε, στον αθλητικό εθελοντισμό από τη μία χώρα στην άλλη και αυτό το οποίο θέλουμε μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών είναι να προωθήσουμε τον εθελοντισμό στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για το ΆΣΕΣ να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για επαγγελματικό, για επαγγελματισμό στον αθλητισμό, δεν μιλάμε για επαγγελματίε αθλητές, μιλάμε για ε, τους πολίτες ε, της ε, Ένωσης που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον, με τον αθλητισμό. Προφανώς, όπως είπε και ο πρόεδρος Ρουπατέλη, αυτή η πρωτοβουλία ε, είναι 10 ετών, είναι μια πρωτοβουλία των, των, των πολιτών που ασχολούνται με τον αθλητισμό προς όφελος των πολιτών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έχουμε την θέληση να, να συνεργαστούμε στενότερα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να δείξουμε κάθε διαφάνεια και όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί ε, αλλά και για όλες μας τις δραστηριότητες ε, στον οικονομικό και δημοσιονομικό τομέα. Ξαναδείω τώρα το λόγο στον πρόεδρο Λουπατέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την φιλοξενία και να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 ε, Νοεμβρίου και σας καλούμε όλους θα δώσουμε την ε, σημαία της πρωτεύουσας ε, του αθλητισμού στην Βαλένθια και θα σας ανακοινώσουμε ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα για τον Αθλητισμό το 2012. Κωνσταντινούπολη, Κάντιθ και αβέρσα είναι τρεις υποψήφιες πόλεις και, στις, ε, και η 30 Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου θα είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική, διότι θα είναι παρούσες και 20 πιο μικρές χώρες που θα δώσουμε και αυτοί. Και σε αυτές μια σημαία είναι ε, πόλεις από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία κτλ. που θα πάρουν και αυτές μια σημαία. Διότι ο αθλητισμό έτσι όπως τον εννοούμε εμεί είναι ένα αθλητισμός φιλία, αδελφόσύνη ανθρωπισμού, ένα αθλητισμός που επιτρέπει την ένταξη των πολιτών της κοινότητας. Ε, προηγουμένως μιλούσατε για τους ε, Ρωμά και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει για να ενταχθούν και τα παιδιά αυτά. Επομένως, εμείς είμαστε στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έτσι ώστε ο αθλητισμός να αποτελέσει ένα πραγματικό κίνητρο και εργαλείο ένταξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ομολογώ πρώτη φορά από εσάς ακούω σήμερα, ίσως και τον Μάρκο όταν μου είπε να μπει το θέμα στη μερίσια διάταξη, μπορούμε να ανοίξουμε κανένα φως. θέλετε Απορώ για το ότι δεν είχαμε ξανακούσει για αυτό το θέμα. Εγώ το 95 ήμουν η πρώτη που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό εδώ μέσα. Κάπου έπρεπε να έχω ακούσει κάτι δεν ξέρω, νομίζω πως δεν είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Α, 2001, ναι. Και από το 2001 έχουν περάσει 9 χρόνια. Κάτι έπρεπε να έχω ακούσει, αλλά ο κύριος Φίσας και ο κύριος Σκουρία από ό,τι φαίνεται ξέρουν αυτό το θέμα. Οπότε χαίρομαι για το ότι θα το συζητήσουμε σήμερα. Θέλω να παρατηρήσω πως το θέμα αθλητισμός και ένταξη νέων στην κοινωνία είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο βεβαίως ε, το λαμβάνουν υπόψη και τα άλλα θεσμικά όργανα. Υπάρχει το Street Football World ε, που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη και προσπαθεί να εντάξει τους νέους μέσω του ποδοσφαίρου. Και βεβαίως ήδη του χρόνου έχουμε το, νέο, το θέμα αυτό των ε, νέων εθελοντών. Οπότε νομίζω πως εδώ πέρα με τη δουλειά σας μπορείτε να βοηθήσετε. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η χρηματοδότηση που έχετε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής και ποια είναι η διάρθρωση που έχετε, πως άνθρωποι βρίσκονται σας στη διοίκηση και πόσους έχετε στη διάθεσή σας για να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε ε, πλην εκτός Βεβαίως ε, πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιος χρηματοδοτεί, αν συμμετέχουν τα κράτη, η πώληση, οι περιφέρειες. Και στο σε αυτό το οποίο λέτε αυτό ισχύει μόνο για το τίλο ή συμμετέχουν και άλλοι ε,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 Γι' αυτό όμως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να ενθαρρύνουμε της, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση, ε, τους δήμους, τις κοινότητες να επενδύσουν στον αθλητισμό. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η οργάνωση είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό, διότι ακριβώς ε, παρουσιάζει μια πρωτοβουλία την οποία μπορούν να εμπνευστούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Υπάρχουν μικρές πόλεις που επενδύουν στον αθλητισμό και αν αυτό τους αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε αυτή η εμπειρία να χρησιμεύσει σαν μοντέλο και για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και για άλλους δήμους και κοινότητες να εμπλακούν στο, με τον, στον αθλητισμό. Διότι στο κάτω-κάτω ό,τι να γίνει εδώ θα πρέπει να γίνει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και λιγότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ παρόμοια άποψη έχω κι εγώ. Και εγώ δυστυχώς παρά το ότι ασχολούμαι αυτά τα θέματα δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικό. Ε, Παρέμεινε κρυμμένο το, πως, το ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του αθλητισμού. Είναι μια πάρα πολύ καλή σκέψη και πολύ καλή ιδέα. Βεβαίω έχει νόημα μόνο αν υπάρχει και μια κάποια δημοσιότητα. και αν υπάρχει μια δημοσιότητα έξω από την ίδια την πόλη βεβαίως. Και δεν έχω αντιληφθεί μέχρι στιγμής πώς είναι η οργάνωση της άξες. Είναι κάποια μέλη, είναι απλοί άνθρωποι, είναι σύνδεσμοι αθλητικοί. Πώς είναι η οργανωτική σας δομή, δεν έχω καταλάβει τίποτα. και να μας πείτε με βάση ποια κριτήρια επιλέγονται μετά οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του αθλητισμού. Eh, eh, Πρέπει να σας πω ότι εγώ ίσως γνωρίζω πιο παλιά αυτή την οργάνωση και ο κύριος Λουπατέλη είναι πάρα πολύ γνωστός και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες για την δέσμευση που έχει αναλάβει και την παρουσία του. Ε, αυτή η οργάνωση, αν θέλετε, δραστηριοποιείται σε τομείς που είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της Λισαβόνας. Ε, μιλάει και το, η συνθήκη της Λισαβόνας για ε, κοινωτικές δραστηριότητες, κοινωτικές πρωτοβουλίες, όμως ε, λαμβάνοντας υπόψη πολύ έντονα το στοιχείο της επικουρικότητας για να αγγίξουμε σαν τον περισσότερους πολίτες. Ε, εδώ ξεκινώντας ε, από αυτήν την οργάνωση ΆΣΕΣ που είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπική αλλά ένα νομικό πρόσωπο ε, και να θεωρήσουμε ότι μπορεί να δραστηριοποιηθούμε, να δραστηριοποιηθεί μάλλον ε, έτσι όπως ε, η Κομισιόν ορίζοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού, την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, υπάρχει μία απόσταση. Θα πρέπει να εξοπλιστούν οι υποψήφιες πόλεις για να... γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μετρήσουμε, αν θέλετε, ε, ας πούμε την, ε, την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στις πόλεις, ε, κατά πόσον αυτές οι εγκαταστάσεις και αυτές οι υποδομές είναι βιώσιμες. Ούτως ή άλλως ε, η Ιταλική Επιτροπή, η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ε, οργάνωση αυτή άσες σαν μια άξια οργάνωση και υπό το φως αυτών των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν ε, και ζητήθηκε η κυρία Πάκ, καλό θα είναι να μας πει η Κομισιόν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κάπως σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας και μέσω της επικουρικότητας με κάποια διαδικασία που θα ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα, ένα label ένα ευρωπαϊκό σήμα σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι μοναδική. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία είναι μοναδική διότι ακριβώς συμμετέχουν πολλές πόλεις και πολλοί πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Λικατέλη και τους συναδέλφους όπως και ο κύριος Φίσας. Είχα και εγώ κάποια επαφή ήδη και αυτά τα οποία άκουσα είναι πάρα πολύ θετικά και ειδικά γνωρίζω πως οι πόλεις οι οποίες θυμήθηκαν το υποδέχτηκαν πάρα πολύ θετικά και υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ε, για διαφορετικές πόλεις, κάτι το οποίο βέβαια είναι σημαντικό γιατί δίνεται έτσι ευκαιρία να αναγνωριστούν έτσι διάφορα πράγματα. και οπωσδήποτε αξίζει να το στηρίξουμε. Τώρα κάνετε κάποιες ερωτήσεις ε, που ήταν σωστές και είμαι σίγουρος ότι θα τις απαντήσει ο κ. Λοκατέλη. Ένας από τους λόγους για τους οποίους βεβαίως φαντάζομαι δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα μέχρι στιγμής είναι πως μόλις τώρα οι αρμοδιότητές μας ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας έτσι αρχίζουν να αναπτύσσονται. Οπότε αναμένουμε φαντάζομαι περισσότερες επαφές εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και να υπάρχει και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη στήριξη από τον λαό για τον αθλητισμό, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε όλα τα θέματα. Αναφέρθηκε λοιπόν, είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να, μπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην οικονομική αξία του αθλητισμού. εγώ μόλις ήρθα από μία συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο για τον αθλητισμό και του είπα πως στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει μια γραμμή του προπολογισμού για τον αθλητισμό. Νομίζω πως ο αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στον αθλητισμό και η πτυχή του εθελοντισμού πρέπει να τονιστεί. Και τέλος να πω πως αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα γίνει τον αριθμό των βουλευτών. Είμαστε πάνω από 100 αυτή τη στιγμή που υπογράφουμε μια δήλωση για τον αθλητισμό και θα ήθελα να σας ζητήσω να υπογράψετε κι εσείς, να το πείτε στους συναδέλφους, να μαζευτούν πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Λουκατέλη που ήρθε και τους συναδέλφους του. Ευχαριστώ, Κορέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση, τη ζητήσαμε γιατί θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει σε σχέση η Ένωση μαζί μας αυτή. Ε, γιατί αυτή η πρωτοβουλία δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστή. Και αυτή η πρωτοβουλία της ΆΣΕΣ είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι υπάρχει αυτή η διαφορά ε, πρωτεύουσα πρωτεύουσες πόλεις και κομοπόλεις αν θέλετε, ε, δημιουργεί μια, μια κίνηση, μεγάλη κινητικότητα, αν θέλετε, αθλητική κινητικότητα σε, στις ε, διάφορες πόλεις, μικρές πόλεις. Άλλο πράγμα η πρωτεύουσα, καλό πράγμα και εκεί, αλλά και στις μικρές πόλεις είναι πάρα πολύ καλό. Ε, και αυτή η ευρωπαϊκή αναγνώριση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες και στις και στις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις ε, πόλεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στους πολίτες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ε, μια προσπάθεια έτσι ώστε παράλληλα με τις ε, πρωτεύουσες, τις αθλητικές πρωτεύουσες, να, μάλλον παράλληλα με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες να έχουμε κάτι και για τον, για τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια κανένα θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει όσον αφορά την χρηματοδότηση διότι δεν, υπάρχει μεγάλη, δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια και θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να εντοπίσουμε κάποια διαθέσιμα κονδύλια. θα ήθελα να ακούσω και την ε, Κομισιόν, παρακαλώ. Ο πρόσωπος Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ καλά είπε ο κύριος ε, Λουπατέλη, ο εκπρόσωπος της ΆΣΕΣ με τον οποίο εδώ και χρόνια έχουμε επαφές, αυτή η πρωτοβουλία της Ένωσης Αθλητικών Πρωτεύουσών υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Αναφέρθηκε και στη Λευκή Βίβλο και αυτό που μπορούμε να πούμε από πλευράς Επιτροπής είναι ότι στο πλαίσιο των περιορισμένων βέβαια δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, Χαιρόμαστε πολύ που μπορούν να υποβληθούν ε, προγράμματα και σχέδια στο πλαίσιο της ε, πρότασης υποβολής προτάσεων και για φέτος και για μελλοντικά χρόνια. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη λευκή αυτή βίβλο και την χάνει της πολιτικής υποστήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής τώρα για τη μελλοντική ανάπτυξη και για τη ε, διαθεσιμότητα πόρων πιστεύω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αξιοποιηθεί ο κοινωτικό προϋπολογισμός και το τι δυνατότητες χρηματοδότησης θα υπάρχουν στον τομέα του αθλητισμού που όπως ξέρετε οι ειδήσει δεν είναι και ιδιαίτερα θετικές δεν είναι ότι πιο ευίωνο θα μπορούσε να περιμένει κανείς αυτόν τον καιρό, αλλά ε, αυτά είχα να πω γενικά εγώ σε εκπρόσωπο της Κομισιόν, αλλά ευχαριστώ να απαντήσω σε τυχόν ειδικέ ερωτήσεις που έχετε. Ωραία, οπότε τελείωσε η συζήτηση. Θα δώσω στον κύριο Λουπατέλη το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα, όσο δυνατόν πιο σύντομα ε, Μπορώ να απαντήσω στα θέματα προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός ε, της, ε, της Ένωσής μας είναι 300.000 ευρώ, ετήσιος προϋπολογισμός. Είχαμε 20.000 ε, από την Ολυμπιακή Ιταλική Επιτροπή, άλλες 100.000 από τα μέλη και άλλες 100.000 από, από ένα κονδύλι που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να επιβιώσουμε διότι είμαστε εθελοντές. Κανείς δεν είναι αμοιβόμενος. Η καρδιά μας χτυπάει γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους Ευρωπαίους πολίτες, κάτι σημαντικό και έχουμε προωθήσει το, την, την, την πρωτοβουλία αυτή λόγω της θελοντικής μας προσφοράς. Και θα συνεχίσουμε διότι θεωρούμε ότι αυτοί οι δήμοι κοινότητες της Ευρώπης αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της αθλητικής πολιτικής, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Και θέλουμε να προωθήσουμε και τις μικρές ε, πόλεις κάτω των 25.000 κατοίκων. Ε, έχουμε μία πρωτεύουσα 9, 9 πόλεις και 19 κομοπόλεις. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε με τη βοήθεια των φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, αν έχουμε και άλλη μία βοήθεια και από πλευράς της Κομισιόν, ακόμα καλύτερα. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Να θέσω ένα ακόμα ερώτημα προς την Κομισιόν. Τα λεφτά τα οποία αναμένεται από εσάς να εγκρίνουμε δηλαδή μπορούν να δοθούν μέσω ενός διαγωνισμού ή όχι. Εάν... Να, να σας ρωτήσω. Δηλαδή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν αναφέρεις τις προπαρασκευαστικές δράσεις στο πλαίσιο του αθλητισμού, ναι, πράγματι το 2009 έγινε μια, είχαμε ένα διαγωνισμό και το 2010 και στο τρίτο έτος των προπαρασκευαστικών δράσεων επίσης ε, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, υποβολή δηλαδή, πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ο προπολογισμό που λέει ο κ. Λουπατέλη προέρχεται από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες εγώ μιλώ ε, για αυτά που είναι αρμοδιότητα της μονάδας για τον αθλητισμό. Ναι, αλλά μπορούν, μπορούν να κάνουν έτσι στην, στην εθελοντική αυτή υπηρεσία. Yeah. Ναι, ναι, δεν ήμουν σαφής. Έχουμε το έτος του εθελοντισμού, νομίζω. Οπότε, πιθανώς ε, μπορεί έτσι να δεν ξέρω, αυτή η εργασία ή όχι. Ναι, πράγματι. Αυτή είναι μια ακόμη δυνατότητα στην προκήρυξη διαγωνισμού για το 2010. Εν ώψη του Ευρωπαϊκού Έτου Εθελοντισμού είχαμε συμπεριλάβει στον τομέα του αθλητισμού ε, τον εθελοντισμό μια από τις Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα προγράμματα ε, υποβάλλεται στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχει και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτου Εθελοντισμού λοιπόν η δυνατότητα, παρότι δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις, να έχουμε δηλαδή πρόσκληση υποβολή προτάσεων. Οπότε ευχαριστώ τους τρεις κυρίους που με πληροφόρησαν για πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Κάποια πράγματα μας ξέφυγαν εδώ πέρα. Αν είναι δυνατόν, και κάθονται εδώ πέρα τρία-τέσσερα άτομα με τον κύριο Κέλλη που είναι πολύ καλά πληροφορημένα. Τώρα λοιπόν τα γνωρίζουμε όλοι όλα. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε να βρείτε χρηματοδότηση και να συνεισφέρει λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσετε τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν τον δρόμο του. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έληξε η σημερινή συνεδρίαση. Τώρα ακολουθεί η συνεδρία των συντονιστών.